Παρακαλώ να σημειώσετε ότι υπάρχει διερμηνία διαθέσιμη σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες της Ένωσης. Είναι ωστόσο απαραίτητο να επιλέξετε το σωστό κανάλι για κάθε γλώσσα. Παρακαλώ λοιπόν να δείτε ποιο είναι το κανάλι της γλώσσας σας. Eh, λοιπόν, ε, με την ιδιότητα τη Πρόεδρου αυτή εδώ τη Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γενικών Ισότητα Άνδρε-Γυναίκε, θα ήθελα να σα πω ότι χαίρομαι που έχω αυτή τη δυνατότητα να σα χαιρετήσω. Χαιρετίζω επίση τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Μπούζεκ, τον οποίο καλωσορίζω εδώ στη συνεδρίασή μα και χαιρόμαστε που ο κύριος Μπούζεκ, ο πρόεδρος, ε, υποσχέθηκε να κάνει μια εισαγωγή για, για να κάνει μια εισαγωγή στην, ε, ε, στον διεθνή Ορτασμό της ημέρας της γυναίκας. Θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε τις απόψεις του Προέδρου κ. Μπούζεκ, κάτι το οποίο είναι ένα, για ένα θέμα το οποίο είναι προσφυλές σε μας και το πώς αντιμετωπίζονται όλα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο γενικότερα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκεκριμένα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, κύριε Μπουζέκ. Thank ε, Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σβένσον, κυρία συνάδελφε. Είναι μια σπουδαία στιγμή σπουδαία μέρα σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μπορούμε να σας φιλοξενήσουμε. Καλώς ορίσατε στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι μια σπουδαία χρονική στιγμή γιατί πριν από 100 χρόνια άλλαξε το ευρωπαϊκό περιβάλλον χάρη στην Ευρωπαϊκή ημέρα τη γυναίκα. Α αρχίσουμε λοιπόν τον εορτασμό από αυτή την συνεδρίαση. Όπω είπε και η κυρία Σβένσον, σε αυτό το κοινοβούλιο έχετε την απόλυτη ποιότητα όσον αφορά την χρήση των γλωσσών σας και υπάρχει απόλυτη ισότητα. Θέλουμε ωστόσο να επικρατήσει και η ισότητα των φίλων δεν είναι τόσο εύκολο όσο είναι με τις γλώσσες. Μπορείτε να ακούσετε αυτή τη στιγμή 23 γλώσσες στην αίθουσα, γι' αυτό και εγώ πια θα μιλήσω πολωνικά. Ας το κάνουμε λοιπόν αυτό, θα μιλήσω πολωνικά, βάλτε τα ακουστικά σας παρακαλώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω την ε, πρόεδρο Φοντέν, την ε, Πρόεδρο Μέρι Ρόμπινσον, αγαπητοί συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα ο κόσμος έχει αλλάξει πολύ από τότε που αρχίσαμε τον εορτασμό της, ε, τον διεθνή εορτασμό της ημέρας της γυναίκας. Μάθαμε πόσο πολύ διώκονται οι γυναίκες και πόσο πολύ στερούνται των βασικών τους δικαιωμάτων. Ωστόσο τα πράγματα έχουν αλλάξει από το παρελθόν, εδώ και 100 χρόνια. Πρέπει αυτό να το αποδεχτούμε, αλλά ξεκολουθούν να υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την επαγγελματική ζωή, τις ε, διάφορες πολιτικές σχετικά με τη γυναίκα υπάρχουν ακόμα ελλείψεις όσον αφορά την ισότητα και τη δικαιοσύνη. Στην ε, αρχικά οι γυναίκες αγωνίζονταν ε, για να έχουν το δικαίωμα να εργαστούν. Τώρα αγωνίζονται για να έχουν το ίδιο, είδος, ε, το ίδιο επίπεδο μισθού για, την, το ίδιο είδος εργασίας, όπως και οι άντρες. Έχουν το δικαίωμα ψήφου, κέρδισαν το δικαίωμα της ψήφου πριν από 100 χρόνια περίπου, αλλά εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις ε, όσον αφορά τη ε, την συμμετοχή τους ε, στα πολιτικά κόμματα και την πολιτική ζωή και γι' αυτό και είμαι υποστηρικτής της εισαγωγής των ποσοστώσεων υπέρ των γυναικών και έχουμε ένα νομοσχέδιο που επεξεργόμαστε στο Βελονικό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή και πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Δεν βλέπω που κάθονται οι Πολωνοί συνάδελφοι. Βλέπω μόνο μία Πολωνή συνάδελφο. Μπορεί να το επιβεβαιώσει φαντάζομαι πόσο μακρύ ήταν ο δρόμος και ο αγώνας για την ισότητα ε, γυναικών και ανδρών. Αλλά είμαστε βέβαιοι πως η κατάσταση θα βελτιωθεί. Το σλόγγαν της σημερινής συνεδρίασης είναι «Οι γυναίκες στην πολιτική». Και γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες στην πολιτική μπορούν να βελτιώσουν το, την κατάσταση των γυναικών γενικότερα, αλλά αυτό που είναι ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι μπορούμε να επηρεάσουμε την εθνική ή την ευρωπαϊκή νομοθεσία με τέτοιο τρόπο, ώστε πραγματικά να αντικατοπτρίζει τις ε, πιο επίγουσες ανάγκες των γυναικών των πολιτών γενικότερα και των γυναικών ειδικότερα, ε, που είναι πολύ πιο ευαίσθητες στις ε, λύσεις και στις ε, απαιτήσει. Είναι πολύ πιο εύκολο όταν υπάρχουν γυναίκες στην πολιτική να βρίσκονται και οι κατάλληλες λύσεις και αυτό έχει αποδειχθεί με πρακτικά παραδείγματα. Η ισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε με την συνυπογραφή της συνθήκης της Ρώμης. Τώρα πια αυτό έχει εγγραφεί και στο θεμελιώδη δικαιώματα, στον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και θα ήθελα να σας δώσω κάποια στατιστικά στοιχεία για το ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Από τη δική μου εμπειρία, όταν γήθηκα της πολωνικής κυβέρνησης, μπορώ να σας πω ότι είχαμε 50 γυναίκες ανάμεσα στις τους ε, αξιωματούχους ε, της ε, κυβέρνησης και των Υπουργείων καθώς και των κεντρικών αρχών. Αυτό το ρεκόρ όμως δεν το έχουμε ακόμα καταρρύψει ήταν ένα απόλυτο ρεκόρ στην πολωνική ιστορία και τώρα ο επικεφαλής ε, του δικού μου γραφείου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένας άνθρωπος που έχει πολύ εξουσία στα χέρια του δηλαδή είναι γυναίκα και ο αριθμός των γυναικών στο δικό μου επιτελείο ανέρχεται στο 54% το Ευρωκοινοβούλιο το ίδιο απασχολεί 60% γυναικών ανάμεσα στους υπαλλήλους του και αυτό που είναι ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι πάνω από το ίμιση των ανθρώπων που έχουν θέσεις που απαιτούν ειδικέ γνώσεις είναι γυναίκες εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Ασχολούνται με πολύ σημαντικά θέματα και λαμβάνουν πολύ σημαντικές αποφάσεις οι γυναίκες εδώ. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσον αφορά τα μέλη του Κοινοβουλίου, του Ευρωβουλευτίνες δηλαδή, είναι 35%. Αυτό βασικά βέβαια εξαρτάται από το ναι, εκλογικό και η νομοθεσία σε κάθε κράτος μέλος. Εγώ θα ήθελα να σας πω λοιπόν ότι Καθώς οι ευρωβουλευτέ εκλέγονται στις χώρες τους, θα ήθελα να σας καλέσω να παρέμβετε ώστε να αλλάξει η εκλογική νομοθεσία με τέτοιο τρόπο ώστε στα τρία χρόνια που θα έχουμε πάλι ευρωεκλογέ να μπορέσουμε να καλωσορίσουμε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο τουλάχιστον 50% γυναίκε. Και αυτό είναι δική σα ευθύνη των εθνικών βουλευτών. Εμεί δεν μπορούμε αυτό να το αλλάξουμε στο Ευρωκοινοβούλιο μόνοι μα Και κάτι ακόμα. Πάνω από 30% γυναίκες λοιπόν στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά όσον αφορά τους ε, ανώτατους ευρωβουλευτές, είναι 40% η εκπροσώπηση των γυναικών, δηλαδή στο Προεδρείο, στο Σώμα των Κοσμητόρων, όσον αφορά τις προεδρίες των κοινοβουλευτικών μας επιτροπών, εκεί εκπροσωπούνται κατά 40%. Τα πιο, πιο σημαντικές θέσεις δηλαδή του Κοινοβουλίου τις κατέχουν κατά 40% οι γυναίκες. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι υπερεκπροσωπούνται οι γυναίκες στο Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί αν δείτε ότι έχουμε 35% ε, γυναίκες ευρωβουλευτίνες αλλά 40% στις ανώτατες θέσεις του Κοινοβουλίου, θα δείτε ότι υπερεκπροσωπούνται. Αλλά αυτό δεν αρκεί γιατί οι στατιστικές δεν ε, μας λένε τα πάντα. Εντάξει, τα πάμε πολύ καλύτερα από το μέσο όρο των Εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρώπης, αλλά ε, δεν είναι και όλα τέλεια. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι σκοπεύουμε και πραγματικά επιθυμούμε να δραστηριοποιήσουμε περισσότερο τις γυναίκες, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για όλους μας αν θέλουμε η Ευρώπη να παίξει καθοριστικό ρόλο σε ολόκληρο τον κόσμο, αν θέλουμε δηλαδή να ε, χειριστούμε, να αντιμετωπίσουμε την κρίση, να αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Θα πρέπει να θυμόμαστε πως οι γυναίκες είναι μητέρες και αν θέλουμε να είμαστε δραστήριες σε, ε, ε, σε επαγγελματικό επίπεδο θα πρέπει να εισαχθεί παντού η μερική απασχόληση, η ευέλικτη απασχόληση, η τηλεεργασία, η πρόνοια για τα παιδιά σε κάθε μεγάλη εταιρεία. Και να εξασφαλίσουμε πως ε, και οι άνδρες θα ασχοληθούν ε, με τη φροντίδα των μικρών παιδιών, γιατί πολύ συχνά ε, οι άνδρες επιθυμούν να ασχοληθούν με τα μικρά τους παιδιά, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό αν θέλουμε να σώσουμε την Ευρώπη από την δημογραφική καταστροφή. Και θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε και τη δουλειά που κάνουν οι γυναίκες ή οι άνδρες στο σπίτι τους όταν έχουν πολλά παιδιά και ασχολούνται με τη φροντίδα τους. Είναι μια πολύ δύσκολη και σημαντική δουλειά αυτή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν δουλεύει μια γυναίκα επειδή ασχολείται με τα παιδιά της. Δουλεύει για το καλό της κοινότητας και μάλιστα κάνει ένα από τα πιο σπουδαιότερα έργα στην κοινωνία. Κάτι ακόμα. Επιχειρήσεις. Πριν από λίγες μέρες μαζί με την Αντιπρόεδρο Επίτροπο Ρέντινγκ δημοσιεύσαμε ένα άρθρο όπου κάνουμε έκκληση στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αυξήσουν εθελοντικά τον αριθμό των γυναικών στα διοικητικά του συμβούλια. Σύμφωνα με τις έρευνες, οι επιχειρήσεις θα έχουν να ωφεληθούν από κάτι τέτοιο, αλλά και εμείς θα ωφεληθούμε από αυτό. Αυτό είναι κάτι ακόμα το οποίο θα πρέπει να αναλάβουμε και να προωθήσουμε. Σε αυτήν την 130η επέτειο της Διεθνούς ημέρας της Γυναίκας, θα ήθελα να συγχαρώ όλες τις γυναίκες γιατί καταφέρατε να επιτύχετε τόσα πολλά τα τελευταία 100 χρόνια και να σας πω ευθέως και σε αυτό απευθύνομαι και στις άνδρες και στις γυναίκες ότι έχουμε ακόμα να αντιμετωπίσουμε μεγάλες προκλήσεις. Δεν υπάρχει ακόμα πλήρης ισότητα στην Ευρώπη και μάλιστα πόρα απέχουμε από την ισότητα εκτός Ευρώπης. Το γνωρίζουμε αυτό πάρα πολύ καλά Πρέπει ακόμα λοιπόν να συνεχίσουμε τη δουλειά για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Να μην ξεχνάμε δηλαδή ότι ενώ γιορτάζουμε την εκατοστή αυτή επέτειο, έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας και εύχομαι κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο. Επίσης να πω ότι ε, κύριε Πρόεδρε, εκ μέρου τη Επιτροπή και όλων των συμμετοχόντων, να σα ευχαριστήσω για αυτήν τη θερμή εισαγωγή εν ώψη τη εορτή τη Διεθνού ημέρα τη εργασία. Και σίγουρα υπάρχουν μεγάλε προκλήσει μπροστά, μα. Αλλά αυτά δεν θα μα απογοητεύσουν ούτε οποιαδήποτε δυσκολία. Εμείς θεωρούμε ότι από κοινού μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα και είμαστε πεπισμένες γι' αυτά. Σας ευχαριστώ πάλι. Λοιπόν, τώρα να σας καλωσορίσω και χαίρομαι που έχουμε εδώ την κυρία Ρόμπινσον, τέος πρόεδρος της Ιρλανδίας, επίσης την κυρία Νικόλ Φοντέν, η οποία υπήρξε πρόεδρος εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευπρόζεκτη και αυτή, επίσης να πω ότι καλωσορίζω όλους συμμετέχοντες, όλες τις συμμετέχουσες από τα Εθνικά Κοινοβούλια και επίσης όσοι είναι παρόντες εδώ από τις υποψήφιες χώρες, επίσης τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι σε αυτήν εδώ τη συνεδρίαση για να έχουμε μια ενδιαφέρουσα ημέρα με όλες τις απόψεις που θα εκφραστούν εδώ και πολλά χρόνια, ξέρετε. Είναι παράδοση το να μαζευόμαστε εδώ με αφορμή τη Διεθνή ημέρα των γυναικών για να ε, ανταλλάξουμε τις εμπειρίες μας, να δούμε ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές κτλ. Και φυσικά να συζητήσουμε τους κοινού μας στόχους και το πώς ακριβώς θα προχωρήσουμε στη δουλειά μας. Φέτος, όπως είπε και ο πρόεδρος κ. Μπούζεκ, είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, διότι επειδή συναντάμε συναντάμε, επειδή φέτος γιορτάζουμε την, έχουμε την επέτειο των 100 ετών από την πρώτη χρονιά που εορτάσει αυτή η μέρα. Χαιρετίζουμε όλους όσοι υπήρξαν ε, πρωτοπόροι πριν από 100 χρόνια και αγωνιστήκαν με θέματα ισότητας και διεκδικήσαν τα δικαιώματα των γυναικών. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό σήμερα να σκεφτούμε σε όλους όσοι πριν από εμά δουλέψανε για αυτά τα θέματα και θα λέγαμε ότι ανοίξανε το δρόμο για αυτές τις διεκδικήσεις και ειλικρινά είναι ευθύνη δική μας εν ε, σε σχέση με αυτούς τους πρωτοπόρους να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες ε, εορτάσει για πρώτη φορά στην Αυστρία, στη Δανία, Γερμανία και στην Αλβετία 19 Μαρτίου του 1911 και πάνω από ένα εκατομμύριο άνδρες και γυναίκες συμμετείχαν στις, στους εορτασμούς εκείνους. Ποια ήταν τα αιτήματα, τα δικαιώματα των γυναικών να δουλέψουν, το δικαίωμα να ψηφίσουν, δικαίωμα στην εκπαίδευση, το δικαίωμα να αναλάβουν κάποια θέση σε δημόσια υπηρεσία. Αυτά ήταν μερικά από τα πρώτα δικαιώματα που διεκδίκησαν οι γυναίκες. Αλλά, αλλά σε λιγότερο από μια εβδομάδα μετά, μετά από αυτή την μαζική θα λέγαμε ε, διεκδίκηση, έγινε κάτι πολύ τραγικό. Πάνω από 140 εργαζόμενες γυναίκες χάσαν τη ζωή τους στο... Σε, μετά την μεγάλη καταστροφή, την πυρκαγιά που έγινε στη Νέα Υόρκη, στο λεγόμενο τρίγωνο της καταστροφής. Πάρα πολλές οι γυναίκες Ιταλικής και Εβραϊκής καταγωγής χάσαν τη ζωή τους. Και αυτό έγινε στη Νέα Υόρκη ακριβώς λίγο μετά την, ε, τον πρώτο εορτασμό τη, για την ημέρα της γυναίκας. Αυτό προκάλεσε μεγάλη ε, προσοχή, ε, δημιούργησε εντύπωση, έσκυψε κανείς πάνω από, τα, από τις συνθήκες κατά τις οποίες δουλεύουν οι γυναίκες και πραγματικά ε, χαρακτήρισε θα λέγαμε και τον εορτασμό, το διεθνή εορτασμό των δικαιωμάτων της γυναίκας. Φέτος τώρα έχουμε ένα θέμα. η θέση των γυναικών στην πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό έχει να κάνει, συνδέεται με τις δικές μας εμπειρίες, την καθημερινή μας ε, δραστηριότητα, ε, με την ιδιότητα το, της πολιτικού, Φερρυπίν, σε καθημερινή βάση, θέματα σε επίπεδο κυβερνητικό στις χώρες μας ή σε ευρωπαϊκό επίσης. Όπως είπε και ο πρόεδρος Μπούζεκ, έχουμε πετύχει κάποια πράγματα. Δηλαδή πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Έχει γίνει πρόοδος παρόλα αυτά είμαστε πεπισμένες και συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας. Υπάρχουν ανισότητες. Τις βλέπουμε. Πρέπει δηλαδή να καταλάβουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Εγώ προσωπικά σκέφτομαι καμιά φορά ότι η εργασία μας όσον αφορά την ισότητα δεν προχωράει και τόσο γρήγορα. Πολύ δύσκολα προχωρούμε. Και τότε συνηθίζω να σκέφτομαι στο εξή ότι υπήρξαν γενναίες ολόκληρες. Κάτω από ποιε προϋποθέσεις μπορούσαν να καθορίσουν τη ζωή τους. Σκέφτομαι τη γιαγιά μου Φερπίν, τη μητέρα μου και συνδέω τη δική μου ζωή, τις προϋποθέσεις που έχω εγώ σε σχέση με αυτές. Αυτό μου δίνει μια εικόνα, καταλαβαίνετε, μια προοπτική. Τι ακριβώς πετύχαμε όλη αυτή τη χρονική περίοδο, σε αυτό το διάστημα. Το σύνολο γυναικών που βλέπουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στα Εθνικά Κοινοβούλιο έχει αυξηθεί. Είναι μια πραγματικότητα. Το βλέπουμε με μια σταθερή ε, μάζουσα τάση τα τελευταία δέκα χρόνια βλέπουμε ένα ποσοστό του 8% σε εθνικά ε, ε, κοινοβούλια και 5% όταν κοιτάμε το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 35,5% συμμετοχής γυναικών με ένα ποσό 35,5 διγενικών ε, σήμερα είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή ποσοστιαίως που έχουμε σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τότε που καθοριστήκαν οι άμεσες εκλογές. Είχαμε μια σταθερή αυξητική τάση μέχρι το 2004, μετά είχαμε μια μικρότερη. Η σημερινή τώρα επιτροπή έχουμε 9 γυναίκες συμπεριλαμβάνει 9 γυναίκες. Ε, και είναι το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είχαμε ποτέ. Τώρα, επίσης, σκέφτομαι και πιστεύω ότι σίγουρα πολλοί συνάδελφοι συμφωνούν και θυμούνται ότι υπήρξαν θετικά αποτελέσματα και ότι πάρα πολλές από εμά συμμετείχαμε σε αυτή τη θετική εξέλιξη τόσο για την ε, παρουσία γυναικών στα Εθνικά Κοινοβούλια όσο και στο Ευρωπαϊκό. και έγινε, ασκήθηκαν πιέσεις και πετύχαμε να έχουμε αυτέ τι περισσότερε συμμετοχέ ε, γυναικών επιτρόπων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2009 μαζευτήκαμε έξω από το Συμβούλιο και εκφράσαμε τις απαιτήσεις μας για τον ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες επιτρόποι. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε την κυρία Ρόμπινσον, η οποία έχει μια ιδιαίτερη θα λέγαμε πολιτική καριέρα, η οποία υπήρξε πρόεδρος, στη χώρα της, στην Ιρλανδία, αλλά η οποία και σε διεθνές επίπεδο υπήρξε στην ύπατη Αρμοσία το ΟΗΕ για ανθρώπινα δικαιώματα και χαιρόμαστε που την έχουμε εδώ μαζί μας. Επίσης θα ακούσουμε μετά τις εμπειρίες της κυρίας Νικόλ Φοντέν η οποία είναι μία από τις λίγες γυναίκες που υπήρξαν πρόεδροι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κυρία Φοντέν έχει δουλέψει επίσης υπουργό στη χώρα της, στη Γαλλία. Μετά, όταν περάσουμε στο δεύτερο μέρος, το πρόγραμμα της ημέρας, τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τις εμπειρίες που έχετε στα Εθνικά Κοινοβούλια, επίσης εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ανταλλάξουμε αυτές τις εμπειρίες μας και να δούμε ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές ούτω ώστε να μπορέσουμε ακόμα καλύτερα να βελτιώσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή. Η εμπειρία των γυναικών πρέπει να ληφθεί υπόψη στην πολιτική ζωή και η συμμετοχή αυτών. Είμαι πεπισμένη ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων όλοι μαζί, όλες μαζί με τις εμπειρίες που έχετε και τις οποίες θα γνωρίσουμε σε λίγο. Τώρα, πριν να δώσω το λόγο στις καλεσμένους μας, θα ήθελα μερικά πρακτικά θέματα να αναφέρω. Σε κάθε θέση υπάρχει ε, ένα έγγραφο στο οποίο μπορείτε να γράψετε αν επιθυμείτε και ομιλίας, ε, αν επιθυμείτε χρόνο ομιλίας. Θα έχουμε δύο μέρη στην στην ε, συζήτησή μας. Το πρώτο θα είναι πιο γενικό και το δεύτερο μέρος του προγράμματος θα δώσει έμφαση στις εμπειρίες και στις πιο καλές πρακτικές. Και εσείς έχετε τη δυνατότητα στο έγγραφο που έχετε εκεί στη, στα σας να, να συμπληρώσετε και να αναφέρετε σε ποιο μέρος από τα δύο της ημέρας στο πρώτο ή στο δεύτερο θέλετε να πάρετε το λόγο. Έχετε όμως τη δυνατότητα, αν το επιθυμείτε, να λάβετε το λόγο και στα δύο μέρη. Αλλά παρακαλώ, αναφέρετε το ρητά στο έγγραφο. Και τέλος, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι τρία λεπτά έχει ο καθένας, η καθεμία στο, στο χρόνο για να μπορέσουν όσο δυνατόν περισσότεροι να έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν. Λοιπόν, άλλη μια φορά καλώς ήρθατε και με μεγάλη μου χαρά θα δώσω το λόγο στην κυρία Μέριν Ρόμπινσον, τέος πρόεδρος στην Ιρλανδία και συνήπατη ορμησία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, πρόεδρος στο Ίδρυμα Μαρή Ρόμπινσον. Καλώς ήρθα λοιπόν και έχετε το λόγο. Thank you, Madam Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, έχω εντυπωσιαστεί μέχρι τώρα με την έντονη έκκληση υπέρ της ισότητας των φύλων από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από εσά κυρία Πρόεδρε. Είναι τιμή για μένα η πρόσκληση να παρουσιάσω την κύρια ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ένα θέμα αγαπητό σε όλους, την πολιτική ενίσχυση και ίση εκπροσώπηση γυναικών σε όλα τα επίπεδα της Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτώντας γύρω μου βλέπω ότι υπάρχει ισορροπία μεταξύ των φύλων και υπάρχουν και υποστηρικτικά άρενα μέλη των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί το θέμα της ισότητας δεν είναι μόνο θέμα των γυναικών, είναι θέμα όλων μας. Και είναι καλό που το βλέπουμε αυτό. Όπως ακούσαμε η εκδήλωση είναι ιδιαίτερη φέτος γιατί γιορτάζουμε την εκατοστή επέτειο της Διεθνούς ημέρας της γυναίκας ε, και γι' αυτό προσεκλήθην στην εκατοστή ε, επέτειο γιατί επίσημα ε, είμαι μέλος των πρεσβυτέρων των Elders που σχηματίστηκε μετά από πρόσκληση του Νέλσον Μαντέλα και Είχα τη δυνατότητα να προσφέρω και νοσηλευτικές υπηρεσίες στους ε, ηλικιωμένους ε, πρεσβυτέρους ε, και πλησίασα λίγο προς τα εκεί. Θα ήθελα να συμβάλλω στην ενθάρρυνση των γυναικών τις επόμενες μέρες να ενώσουν τα χέρια με τις αδελφές μας όλο τον κόσμο. Πέρσι στις 8 Μαρτίου και εγώ ενώθηκα με εκατοντάδες γυναικών και ορισμένων ανδρών που υποστήριζαν καθώς ε, περπατήσαμε στη γέφυρα του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη ε, ενωμένοι με χιλιάδες γυναίκες πάνω σε άλλες γέφυρες, <clears throat> σε 100 πόλεις και άλλα μέρη σε όλο τον κόσμο. Αυτή η εκδήλωση οργανώθηκε από τη Ζαϊνή Ψαλμπή, από τις γυναίκες για τη Διεθνή των Γυναικών και άλλες ε, διεθνείς οργανώσεις, μη κυβερνητικέ οργανώσεις και θέλουν να ενώσουν περισσότερες γυναίκες και άνδρες 8 Μαρτίου φέτος σε γέφυρες. Ελπίζω ότι κάποια μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, στην Ευρώπη θα μπορέσουν να βρουν μια γέφυρα για να πραγματήσουν την επόμενη Τρίτη μαζί με άλλους, τραγουδώντας μάλιστα. Η εκατοστή επέτειος είναι μια χρονική στιγμή που μας επιτρέπει να σκεφτούμε το παρελθόν και το, να σχεδιάσουμε το μέλλον. Το 93. Είχα την τιμή να επισκεφθώ ε, τη Νέα Ζηλανδία διότι εόρταζε η χώρα εκείνη το γεγονός ότι ήταν η πρώτη παγκοσμίως που έδωσε ψήφο στις γυναίκες το 1893. Ε, χαίρομαι που μπορώ να πω και περηφανεύομαι για το γεγονός ότι άρχισε η νομοθεσία και η νομοθετική προσπάθεια από έναν Ιρλανδό, τον Τζον Μπάλανς από το Άλστερ. Η πραγματική δύναμη ήρθε από τις γυναίκες της Νέας Ζηλανδίας που ε, πάνω στα ποδήλατα κάλυψαν εκατοντάδες βίλια σε ορεινές περιοχές ε, στα δύο νησιά συλλέγοντας υπογραφές. Γνωρίζομαι τους αγώνες για την εξασφάλιση δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες στις διάφορες χώρες στην αρχή του 20ου αιώνα και αργότερα για τον αγώνα για να μπορούν να εκλέγονται βουλευτίνες. Σε κάποια μέρη του κόσμου αυτοί οι αγώνες είναι πρόσφατοι και συνεχιζόμενοι. Οι γυναίκες στο Κουβέιτ ε, το 2005 πήραν δικαίωμα ψήφου και στις αραβικές περιοχές συνεχίζουν να παλεύουν για να θέτουν υποψηφιότητα στο κοινοβούλιο, να γίνονται υπουργοί. Ιδιαίτερα νέες γυναίκες, γι' αυτό είναι αξιοσημείωτο, κατέβηκαν στους δρόμους ε, πρόσφατα στις αραβικές χώρες παρά τη βία που ασκείται εναντίον τους, ζητώντας μεγαλύτερες ελευθερίες, συμμετοχή, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Αυτό το λαϊκό κίνημα που διαφοροποιείται σε κάθε χώρα θα μπορούσε να δράσει μετασχηματιστικά αν οι γυναίκες μπορέσουν να συμμετέχουν πλήρως και ισότιμα στις ε, νέες, ε, στα νέα νομικά και συνταγματικά μορφώματα στην την Ισία, Αίγυπτο, Μπαχραήν, Λιβύη και αλλού. Είναι πολύ σημαντική η εξουσία των γυναικών και ε, για τη δημοκρατική ανάπτυξη στον αραβικό κόσμο διότι όταν οι γυναίκες μπορούν να συμμετέχουν στο κοινοβούλιο θέτουν θέματα που άλλοι τα ε, παραγνωρίζουν. Ε, όταν υπάρχει μια κρίσιμη μάζα γυναικών μελών αλλάζουν τις προτεραιότητες. Η συμμετοχή των γυναικών στην κυβέρνηση τις κάνει πιο αντιπροσωπευτικές, ε, πιο υπόλογες, υπεύθυνε και ξεπερνούν ευκολότερα οι γυναίκες στις εθνοτικές, φιλετικές και θρησκευτικές διαφορές. Και να μην συγχαίουμε τις έννοιες άραβας και ε, μουσουλμάνος, Ισλάμ και αραβικός κόσμος. Ε, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσουν το μετασχηματισμό στη δημοκρατία στον αραβικό κόσμο. Είναι προς όλων, τον το συμφέρον αυτό ε, είναι σημαντική τάση σήμερα στην Ευρώπη προς μια Ισλαμοφοβία η οποία βεβαίως ε, γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης μακροπρόθεσμα. Ε, θα πρέπει να ε, μην έχουμε Ισλαμικές, Ισλαμίστριες, Φεμινίστριες όπως δεν έχουμε Εβραίες ή Χριστιανές Πιστεύω ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα οι γυναίκες μέλη του Κοινοβουλίου θα πρέπει να παίξουν ρόλο. Ε, η, ε, ε, όπως είπα σε μια διάσκεψη στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα παρουσιάζονται ε, αυτές οι ε, ορισμένες αντιδραστικές κινήσεις. Πάντως θεωρώ ότι πολλά μπορούν να γίνουν στις ευρωπαϊκές εκλογικές περιφέρειες και στον αραβικό κόσμο υπέρ των γυναικών. Υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, μπορεί να λάβουν χώρα βραχυπρόθεσμα σχετικά. Ε, έχω γίνει αισιόδοξη έχοντας δει το μετασχηματισμό σε δύο χώρες, τη Ρουάντα και τη Λιβερία. Ήμουν η πρώτη αρχηγός κράτους που πήγα στη Ρουάντα μετά την γενοκτονία των 90 και επέστρεψα εκεί το 95 για να ενημερώσω για τα δεινά του λαού της Ρουάντας στα τα, τα Ηνωμένα Έθνη. Ε, είναι τρομερή η συνέπεια μιας γενοκτονίας. Ε, οι γυναίκες ήταν γεμάτες ανθρώπινα οστά, ε, δέματα με ρούχα και παπούτσια, πολλά ανήκαν σε παιδιά που είχαν σφαγεί. Αλλά ε, πέρα από αυτή τη φρίκη υπήρχαν και ωραίες εικόνες. Ε, σε πολλές από τις εκκλησίες ε, και γύρω στο γύρο χώρο άνθιζαν λουλούδια με τα ωραιότερα χρώματα, ροζ, κόκκινα, κάποια εκπρόσωπος μη κυβερνητικής οργάνωσης μου είπε ότι άνθησαν τόσο πολύ γιατί το χώμα είχε ποτιστεί με αίμα. Τη τρίτη μου επίσκεψη στη Ρουάντα ως πρόεδρος έλαβε χώρα το Μάρτιο του 1997 για να συμμετάσχω σε μια παναφρικανική διάσκεψη γυναικών στο Κιγκάλι που οργανώθηκε από χείρες εν που επιβίωσαν και αντιμετώπισαν το τραύμα τους. Αυτή η διάσκεψη έβαλε τη Ρουάντα σε ένα δρόμο ε, ανάληψης δέσμευσης για να ενισχύσει τις γυναίκες σε κάθε επίπεδο να αντιμετωπίσει ε, νομοθεσίες που οδηγούσαν σε διακρίσεις ε, νόμοι για τη γη, για το κληρονομικό δίκαιο να δώσει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν, να εκπαιδευτούν και πραγματικά έτσι ε, αυξήθηκε και το ποσοστό των γυναικών βουλευτών. Ε, μπόρεσαν λοιπόν τα λουλούδια να ανθίσουν πάλι. Ο μετασχηματισμός της Λιβερίας άρχισε με τις ακτιβίστριες εκεί που ε, αδειμονούσαν για τον αργό ρυθμό των ειρηνευτικών συνομιλιών που διεξήγαγαν οι άνδρες. Τους πλαισίωσαν στο χώρο που έγινόντουσαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Ε, αυτό το κάλυψε και σε ένα ντοκιμαντέρι Άμπι Disney να γυρίσει ο διάβολος στην κόλαση. Οι εκλογέ εκεί το 2005 ε, οδήγησαν στην εκλογή της πρώτης προέδρου αφρικανικής χώρας της Έλεν Τζόνσον Τσίρλιφ και ε, οι γυναίκες της Λιβερίας ε, μπόρεσαν να αξιοποιήσουν και το ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια σαν οργανωτικό εργαλείο. Ε, μια διεθνής διάσκεψη στη Λιβερία 8-9 Μαρτίου 2009 ε, που συνδιοργανώθηκε από τις Προέδρους Λιβερίας και Φιλανδίας εόρτασε την πρόοδο. Η Μισελ Μπασλέ, εκτελεστική διευθύντρια, του πρόσφατα ε, δημιουργημένου φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες επέλεξε να πάει στη Μονοροβία για την πρώτη Διεθνή ημέρα της γυναίκας ε, αναγνωρίζοντας ότι η Λιβερία ε, ενισχύει τις γυναίκες υπό την πρόεδρό της. Και έτσι περνώ σε ένα άρθρο που συνέγραψα πριν από λίγο καιρό με τον Κόφι Ανάντζη Μικάρτερ και Γκράσα Μασέλ ω μέλο των Πρεσβυτέρων μια ομάδα που συνεκλήθη μετά από έμπνευση την Έλσον Μαντέλα και υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Ντέσμον Τούτου ε, μπορούμε να, ε, θέλουμε να επανεπιβεβαιώσουμε τη σημασία της προώθησης του ηγετικού ρόλου των γυναικών. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι σήμερα ένα αυξανόμενος αριθμό γυναικών έχουν αξιώματα με πολιτική επιρροή σε όλο τον κόσμο, αλλά για μέτρα τα εκατομμύρια γυναικών και κοριτσιών λίγα μπορούμε να, κάνουμε, λίγα μπορούμε να γιορτάσουμε. Οι καταστάσεις που αντιμετωπίζουν είναι πραγματικά αφόρητες. Οι γυναίκες είναι οι περισσότερες από τους, από τους του κόσμου. Ε, βία ε, με βάση το φύλλο, συστηματικές διακρίσεις ενάντια στις γυναίκες συνεχίζονται σε πολλέ χώρε του κόσμου. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα κίνδυνο σε περιοχές συγκρούσεων, η θνησιμότητα των ε, μητέρων, ε, η προσβολή από HIV και AIDS στις γυναίκες ε, επιδεινώνεται. Οι έφηβες γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες νέες γυναίκες πολλές φορές ε, λησμονούνται στις προσπάθειες βοήθησης των φτωχών κοινοτήτων. Δυστυχώς αυτές οι ανησυχίες θα συνεχιστούν για πολλά χρόνια ακόμα, αλλά ξέρω ότι αντιμετωπίζονται στη Μονροβία ε, τώρα. τι γίνεται λοιπόν με την ενίσχυση, την πολιτική ενίσχυση των γυναικών στις ευρωπαϊκές χώρες. Βέβαια, σημειώθηκε σταθερή πρόοδο στι τελευταίε δεκαετίες σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για την ίση μεταχείριση, με σημαντικέ υποθέσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και των Εθνικών Δικαστηρίων, πρωτοβουλειών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλω να αποτύσω φορό τιμή στο έργο τη Επιτροπή Γυναικών και σε εσά, κυρία Πρόεδρε. Ε, οι εκθέσει σχετικά με την ισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2010 εξετάζει πολλέ προηγούμενε πρωτοβουλίε, συμπεριλαμβάνοντα το ψήφισμα από το 13 Μαρτίου 2007 για τον ε, οδικό χάρτη για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 2006-2010. Στην έκθεση παρουσιάζονται 26 σημεία. Τα πρώτα 14 αναφέρονται σε θέματα απασχόλησης ε, γυναικών, ισότητας γυναικών, ε, στην αμοιβή, στι συνθήκε εργασία. Το σημείο 15 όμως είναι λίγο αδύναμο και παραθέτω. Χαιρετίζει τι προσπάθειε που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική. Ε, τάσεται λοιπόν υπέρ τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ειδικότερα σε θέσει ευθύνη τονίζει όμως ότι περαιτέρω προσπάθειες θα πρέπει να αναλυφθούν σε εθνικό, περιφερειακό και ε, τοπικό επίπεδο. Η έκθεση αναφέρει ότι μόνο 3% των μεγάλων επιχειρήσεων ε, έχουν πρόεδρο γυναίκα και καλεί τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσέξουν ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες γυναικών, ειδικότερα γυναίκες με αναπηρία και γυναίκες Ρωμά. Ε, διαβάζοντας την έκθεση, κυρία Πρόεδρε, ε, θεώρησα ότι ήταν σαν ένα εγχείρημα όπου έπρεπε να ε, πατηθούν τα σωστά κουμπιά. Ε, και αυτό έγινε. Υιοθετήθηκε από 22 ψήφους υπέρ 2 κατά και θεωρώ ότι νομίζω ότι θα υποβληθεί στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα. Να συνοψίσω την αξία της εκπροσώπησης γυναικών παραθέτοντας ένα εδάφιο από μια πρόσφατη έκθεση του NDI, του Εθνικού Δημοκρατικού Ινστιτούτου για τη Δημοκρατία και τις Προκλήσεις για Αλλαγή ε, ένας οδηγός. Η έκθεση ε, παρουσιάζει ε, μελέτες περιπτώσεων σε όλο τον κόσμο, τη μακρά εμπειρία που υπάρχει και θα το θέμα ως εξής η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική βοηθεί ε, στην επίτευξη της ισότητας μεταξύ των φύλων, ε, επηρεάζει όλα τα πολιτικά θέματα που εξετάζονται, όλες τις λύσεις που προτείνονται. Πολλά δείχνουν ότι εάν περισσότερες, καθώς περισσότερες γυναίκες ε, προβάλλονται σε εκλόγιμες θέσεις θα αυξάνονται ε, τα ε, πολιτικά θέματα που επιλύονται, οι προτεραιότητες που θα γίνονται πιο σωστές για τις οικογένειες, τις γυναίκες, τις ε, φιλετικές μειονότητες. Είναι πολύ σημαντικό για τη δημοκρατία γενικότερα αυτό όταν οι γυναίκες είναι πολιτικές, πολιτικοί ηγέτες αυξάνεται το επίπεδο ζωής είναι θετικέ οι εξελίξει. Η παρουσία των γυναικών στην πολιτική διασφαλίζει ότι εκπροσωπούνται τα προβλήματα των γυναικών και άλλων περιθωριακών ομάδων. Η ηγετική θέση των γυναικών, το ύφο του στην επίλυση των κρίσεων ε, στηρίζεται στα δημοκρατικά ιδεώδη. Ε, είναι πολύ πιο ε, συνεργάσιμες και ακολουθούν λιγότερο στιγνά την ιεραρχία οι γυναίκες. Επίσης δουλεύουν λιγότερο κομματικά, περισσότερο διακομματικά. Επίσης οι γυναίκες νομοθέτες βλέπουν την κυβέρνηση ως ένα εργαλείο να ε, βοηθήσουν ε, μειονοτικές ομάδες. Ε, οι γυναίκες επίσης είναι αφοσιωμένες στην ειρήνη, την οικοδόμηση της ειρήνης, την ανασυγκρότηση μετά από συγκρούσεις. Οι γυναίκες δυσανάλογα υποφέρουν σε ένοπλες συγκρούσεις και συχνά τάσσονται πιο στεναρά υπέρ της σταθεροποίησης, ανασυγκρότησης και της πρόληψης περαιτέρω συγκρούσεων για να αντιμετωπίσουμε τα παγκόσμια προβλήματα και τους στόχους ε, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες, να τους δώσουμε ε, ε, εξουσία και να τις στηρίξουμε στις ηγετικές τους θέσεις. Γιατί όμως η συμμετοχή των γυναικών στο πολιτικό επίπεδο στην Ευρώπη, αφού έτσι είναι τα πράγματα, αντιμετωπίζει προβλήματα. Ε, Σημερίζομαι την αισιοδοξία του Προέδρου, αλλά ενώ 10 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πάνω από 27% εκπροσώπηση των γυναικών στην κάτω βουλή, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με επικεφαλή στη Σουηδία που είναι 45%, η πλειοψηφία συμπεριλαμβάνοντας και τη δική μου χώρα είναι κάτω από το 23% και δύο χώρες έχουν γυναίκες σε ποσοστό κάτω από 10%. Οι παραδοσιακοί φραγμοί παραμένουν αρκετά ισχυροί και αποτρέπουν τις γυναίκες υποψήφιες. Ε, δεν υπάρχουν αρκετοί οικονομικοί οικονομικοί πόροι, είναι δυσανάλογε οικογενειακέ υποχρεώσει, υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον, ε, μια προτεραιότητα πολλών, προτίμηση πολλών γυναικών να λειτουργήσουν στην κοινωνία των πολιτών γιατί είναι πιο φιλικό το περιβάλλον. Η κάλυψη των ε, ΜΜΕ, των αποφάσεων ε, του πρόσφατου παρελθόντο των Λύσια Ροντσούλη και Ρασιντάντα μελών του Κοινοβουλίου, τότε δείχνουν πώς πραγματικά είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην ε, ε, οικογενειακή και πολιτική ζωή τους οι γυναίκες. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια αυτής της εκατοστής επαιτίου, θα πρέπει να ρωτήσουμε, εμείς στην Ευρώπη είμαστε έτοιμοι πραγματικά να καταπιαστούμε με αυτά τα προσκόμματα ε, και τα εμπόδια μέσα σε μία δεκαετή περίοδο μετασχηματισμού. Οι χώρες είναι έτοιμες να εισαγάγουν εθνικές ποσοστώσεις για τις εκλογές τοπικές και βουλευτικές για να διορθωθούν οι ενισορροπίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εθνικές κυβερνήσεις είναι έτοιμες να παράσχουν οικονομικούς πόρους για να εκπαιδευτούν, να εξοπλιστούν οι υποψήφιες γυναίκες σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα εθνικά κοινοβούλια προτίθενται να προσαρμόσουν τις διαδικασίες τους για να επιτρέψουν στις γυναίκες μέλη τους να έχουν καλύτερη ισορροπία ζωής και δουλειάς. Τα πολιτικά κόμματα στις ευρωπαϊκές χώρες ενδιαφέρονται να διερευνήσουν πώς θα αλλάξουν το ανδροκρατούμενο ήθος τους για να προσελκύσουν γυναίκες μέλη. Οι γυναίκες είναι έτοιμες να δεχτούν την ευθύνη της ανάληψης ηγετικών θέσεων και να δώσουν ένα όραμα για το πώς θα, πλησιάσει, πώς θα ε, κλείσει το δημοκρατικό ε, έλλειμμα στην Ευρώπη σήμερα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα και το ευρύτερο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και κλιματικό περιβάλλον και οι προκλήσεις σε όλα αυτά τα επίπεδα ε, προϋποθέτουν ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ε, δεχτεί ένεση από νέο αίμα ζωντάνια από τις γυναίκες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι αλλά και ρεαλιστές ταυτόχρονα. Το 2008 η Επιτροπή του Ηνωμένου Βασιλείου για την Ισότητα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δημοσίευσε μια έκθεση ε, φίλο και εξουσία» και μεταξύ άλλων αναφέρει και παραθέτω «Ένας αλιγκάριθ μπορεί να συρθεί καθόλου το μήκος του κινέζικου τείχους σε 212 χρόνια». Ε, χρειάζεται λίγο παραπάνω από τα 200 χρόνια που θα χρειαστούν για ίση εκπροσώπηση στο Κοινοβούλιο των γυναικών. Δεν θέλουμε μικρές αυξήσεις. Δεν θέλουμε ταχύτητα του σαλιγκαριού. Θέλουμε ε, αλλαγές που θα μετασχηματίσουν την κοινωνία αν πρόκειται να, αναφερθούμε, να ασχοληθούμε αποτελεσματικά με τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ρόμπινσον. Και τώρα αμέσως θα δώσω το λόγο στην κυρία Φοντέν, παρακαλώ. Χαίρομαι πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, που θέλατε να με ε, συμπεριλάβετε σε αυτή την ε, συνεδρίασή σας που γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από την πρώτη, πρώτο της ε, ημέρας της γυναίκας. Είναι μια ευκαιρία να δούμε ποιες είναι ε, ποια είναι η πρόδοση η οποία υπετέφθηκε. Ο αγώνας όμως παραμένει ακόμα σαν ένας αγώνας για την ισότητα ανδρών γυναικών και δει σε επίπεδο πολιτικό γιατί είναι και το θέμα το οποίο έχετε επιλέξει. Σα συγχαίρω που θέλατε να συμμεριλάβατε σε αυτή τη συνεδρίαση, στη συνάντηση με τα μέλη το, από τα Εθνικά Κοινοβούλια, καθώς και από τις, χώρες, τις υποψήφιες χώρες. Τα 23 χρόνια που είμαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μου επιτρέψαν να καταλάβω τον κοινό ρόλο που έχουμε εμείς από τα Εθνικά Κοινοβούλια με ε, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μπορέσουμε να καλύψουμε, να ξεπεράσουμε αυτό που λέμε έλλειμμα Ο, δημοκρατικό. Όταν ήμουν αντιπρόεδρος στο Κοινοβούλιο σε σχέση με, και ανέλαβα τις σχέσεις ανάμεσα στις, στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έκανα μεγάλη προσπάθεια και με θέρμη αντιμετώπισα αυτά τα θέματα. Η πρώτη μου παρατήρηση θέλει να υπογραμμίσει την αποφασιστικότητα που είχαν πάντα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προχωρήσει αυτό το θέμα ε, με τις διακρίσεις βάρους των γυναικών. Όχι μόνο γιατί είναι θέμα ισότητας, δικαιοσύνης, αλλά διότι έχει να κάνει και με την λειτουργία της δημοκρατίας αυτή τη θεμελιώδη θα λέγαμε αξία για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση και για τη σωστή εναρμόνιση των κοινωνιών μας. Επίσης έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα με την βασική αρχή που εντάσσεται στη συνθήκη της Ρώμης και όπου υπήρχαν μεγάλες ε, αντιδράσεις και επιφυλάξεις από τις χώρες μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να χαιρετιστεί με την πρωτοβουλία που παίρνει. Επίσης όμως η προσπάθεια δυναμική του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου και δι της Επιτροπής των Γενικών που δημιουργήθηκε το 1984 και όπου φυσικά και εγώ αμέσως θέλησα να συμμετάσχω. Η ουσιαστική πρόδρος που επιτεύχθηκε έγινε χάση στην κοινή αυτή ε, δράση. Κανένας δεν αφιβάλλει και, και μπορεί να μας το επαληθεύσουν εδώ ε, οι συμμετέχοντες ότι δημιουργούν παρόλα αυτά όλες τις προσπάθειες μια νέα δυναμική η οποία είναι απαραίτητη διότι σήμερα θα διαψώνουμε τα Σίγουρα έχει γίνει πρόοδος αλλά έχουμε μια, ένα απολογισμό ο οποίος δεν είναι αυτός που θα επιθυμούσουμε και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Σε σχέση με αυτό, στα έξι λεπτά που έχω στη διάθεσή μου θα ήθελα να κάνω κάποιες νήξεις. Πρώτον, καταρχήν, να πω ότι επιθυμώ να... το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι παραδειγματικό, να είναι δηλαδή η αιχμή του δόρατος αυτόν τον αγώνα. Τόσο στο σχετισμό ανδρών-γυναικών, αναφέρθηκε αυτό επανειμένο, 35,5% σήμερα, πολύ ανώτερο από ό,τι βλέπουμε στα περισσότερα εθνικά κοινοβούλια με μέσο όρο 24%. Επίσης το θέμα του καταμερισμού των αρμιδοτήτων στα διάφορα όργανα, προέδρους, αντιπροέδρους, προέδρους επιτροπών. Αλλά παρόλα αυτά παραμένουν πολλά πράγματα τα πρέπει να γίνουν όσον αφορά τα προεδρία των πολιτικών ομάδων. Τον Ιούλιο του 1999 όταν ε, εξελέχθη πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο λυπόμουνα που έπρεπε να περιμένουμε 20 χρόνια μετά από την εκλογή της Σίμων Βέιλ για να έχουμε ξανά μια γυναίκα πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω αυτό να μην ξαναχρειαστεί να γίνει, να μην περιμένουμε δηλαδή άλλα τόσα 20 χρόνια. Τέλος, όταν σε αυτό εδώ το ημικύκλο θίγονται τα μεγάλα κοινωνικά θέματα και τα πιο ευαίσθητα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει πάντοτε να είναι σε επιφύλαξη να μπορεί να ε, υποστηρίζει τα όσα έχουν διεκδικηθεί και δεν θα πρέπει όμως να δράσει μόνο. Θα πρέπει να δούμε και τις κυβερνήσεις, τις εθνικές, τα πολιτικά κόμματα, όλοι μαζί να κινητοποιηθούν ώστε να μπορέσει να υποστηριχθούν τα θέματα των γυναικών στην πολιτική. Ξέρω, υπάρχει μια αμφισβήτηση όσον αφορά το θέμα της ποσόστοσης. Κι όμως έχουμε δει ότι με μια ρύθμιση περιοριστική ε, που έχει γίνει, η ισότητα ανθρώπων γυναικών μπορεί να ε, βελτιωθεί και να βελτιώσει την κατάσταση. 6 Ιουνίου 2000 είχαμε ένα νόμο στη Γαλλία όπου αναφέρεται η ισότητα ανθρώπων γυναικών για τις περιφερειακές και περιφερειακές ε, εκλογές αλλά καθώς και σε επίπεδο εθνικών εκλογών και ευρωπαϊκών. Σήμερα τι διαπιστώνουμε ότι αυτός ο νόμος προκάλεσε μια επανάσταση τόσο σε τοπικό επίπεδο όπου η πολιτική είναι πιο κοντά στον πολίτη παρόλο που στην πραγματικότητα ε, η συμμετοχή γυναικών στα περιφερειακά συμβούλια είναι 35% κυρίως οι, οι λίστες, ε, στις λίστες έχουμε επικράτηση των ανδρών και βλέπουμε ότι τα πολιτικά κόμματα ακόμα προτιμούν αντί να σεβαστούν την ισότητα, δίνουν μια προτεραιότητα στου άνδρε. Αλλά σε γενικέ γραμμέ ο απολογισμό είναι θετικό. Θα πρέπει να συνεχίσουμε και να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Επίση, οι εθνικέ κυβερνήσει θα πρέπει να ανησυχήσουν λίγο, να ασχοληθούν, να εξασφαλίσουν μέσα, ούτω ώστε να παροτρύνουν τι γυναίκε να μπουν στον πολιτικό σύμβο. Σε πολλέ από τι χώρε μα, και στη δική μου συγκεκριμένα, η πολιτική έχει χάσει την αξιοπιστία της και επιβάλλεται ώστε να γίνει μια προσπάθεια ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία της στα μάτια του πολίτη, του μέσου πολίτη. Επίσης να προσθέσω δύο προβληματισμούς που αποφθύνονται στις γυναίκες. Στο πολιτικό περιβάλλον, όπως και αλλού, η γυναίκα θα πρέπει να αποδείξει τις ικανότητες της. Είναι καταδικασμένη τρόπον την να διαπρέψει το ξέρει όμως αυτό. Και το θεωρεί μάλλον ένα κίνητρο. Θα πρέπει παρόλο από τη μια να κρατήσει τη θηλυκότητά της, αλλά παρόλα αυτά να προσπαθήσει να επιβληθεί αντί να περιμένει να έρθουν να τη βρουν. Και τέλος, η γυναίκα η οποία περνάει σε ένα σημαντικό πόστο πολιτικό θα πρέπει να είναι σε επιφύλαξη. Θα πρέπει να αποφύγει τις παγίδες, θα πρέπει να προσέξει στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται και η θέση της είναι πάντοτε σε κρίσιμη θα έλεγα. Θα πρέπει να το επαναλάβουμε αυτό επανελειμμένα. Και εγώ από τη δική μου πλευρά το έχω ζήσει αυτό εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δει κατά την περίοδο που εξελέχθη πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αναφέρθηκε σε αλληλεγγύη ο κύριος πρόεδρο Μπούζεκ. Αυτή η αλληλεγγύη επιτρέπει στη γυναίκα να προχωρήσει και να βελτιωθεί η, σχέση, η θέση μάλλον των γυναικών στον πολιτικό στίβο. Επίσης να πω, επίσης να αναφερθώ στην εμπειρία της χώρας μου. Το 1974, 70% των Γάλλων λέγανε δεν θα επιθυμούσαν μια γυναίκα πρόεδρο της Γαλλίας. Σήμερα τι βλέπουμε όλα δείχνουν ότι 90% θα δεχόντουσαν χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς επιφύλαξη, όπως είναι το ίδιο που βλέπουμε και στη Γερμανία, στη Λιθουανία, όπου έχουμε καγκελάριο, πρόεδρο κτλ. Λοιπόν, αυτά ίσως για τη Γαλλία για το 2012. Βλέπουμε δηλαδή η νοοτροπία έχει αλλάξει και αυτό είναι ελπιδοφόρο. Θα πρέπει να την ενισχύσουμε αυτή τη τάση, να τη βοηθήσουμε, να τη διευρύνουμε. Και δεν αμφιβάλλω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γενικών και την Ισότητα των ε, Φίλων θα συνεχίσει να υποστηρίζει αυτό το θέμα και θα συμβάλλει τα μέγιστα. Επι... Ε, θα ήθελα να ευχηθώ λοιπόν σε αυτή την επέτειο ό,τι καλύτερο για την επέτειο της ημέρας της γυναίκας και είμαι πεπισμένη ότι με το ταλέντο της και το κουράγιο της η γυναίκα θα πετύχει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Ρόμπισον, επίσης την κυρία Φοντέν. Νομίζω ότι είχαμε μια καλή γενική ε, εικόνα για το τι υπήρξε πετυχημένο για τις γυναίκες, αλλά και ποιες είναι οι προκλήσεις του μέλλοντος. Και κυρίως τίθεται το θέμα να προβάλλουμε κάποια ερωτήματα όπως είπε η κυρία Ρόμπινσον ότι η Ευρώπη φέρει μέσα σε 10 χρόνια επιθυμεί, ίσως θα πρέπει να πετύχει ε, ισότητα στη συμμετοχή ανδρών, ανδρών γυναικών στην πολιτική αλλά και σε άλλους τομείς. Είναι ε, ερωτήματα τα οποία θα δούμε εδώ κατά τη διάρκεια της ε, συνεδρίασης και Επίσης, ε, αναφερόμενο στην παρουσίαση της κυρίας Φοντέν για την αλληλεγγύη ανάμεσα στις γυναίκες είναι σημαντική και είναι σημαντικό λοιπόν να συμβάλλουμε, να παροτρύνουμε, να ενθαρρύνουμε μια γυναίκα όταν αναλαμβάνει ένα δημόσιο, δημόσιο αξίωμα και είναι καλό να γίνει αυτό όλο και περισσότερο και να αισθάνεται μια γυναίκα ότι έχει στήριξη σε αυτήν εδώ την προσπάθεια ούτως ώστε δηλαδή στο τέλο να μην καταλήξει μια, ένα, το, η κατάληψη ενό πόστου από μια γυναίκα το άλοθη στην πολιτική ζωή. Ευχαριστώ λοιπόν ξανά τις κυρίες για την εισαγωγή που κάνανε. Τώρα μπορούμε να περάσουμε σε ένα διάλογο και να υπενθυμίσω ότι το πολύ τρία λεπτά θα έχει κάθε ομιλητή ομιλήτρια στη διάθεσή του, διότι είναι πολλοί οι οποίοι και πολλέ που θέλουν να παρέμβουν. το πρώτο όνομα, η κυρία Φιγκερίδο είναι στο κατάλογο μιλητών, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο μέλος. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Eh, eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ όλες τις γυναίκες που είναι σήμερα παρούσες αλλά και τις, όλες τις ευρωπαίες γυναίκες αλλά και τις γυναίκες ολόκληρο τον κόσμο κυρίως αυτές που σήμερα υποφέρουν στις χώρες τους γιατί υπόκειται σε διακρίσεις ή αγωνίζονται για την ελευθερία όπως βλέπουμε να γίνεται σε πολλές και διάφορες χώρες ή γίνονται θύματα πολέμου ε, αγωνίζονται για την ειρήνη όλες τις γυναίκες λοιπόν από εδώ ένας χαιρετισμό ιδιαίτερος για τις γυναίκες που εξακολουθούν να υποφέρουν και που εξακολουθούν να αγωνίζονται και προσπαθούν να πετύχουν ε, την ισότητα, τα δικαιώματά τους, ευκαιρίες για τις ίδιες αλλά και να μπορέσουν να καθορίσουν το ίδιο τους το πρόγραμμα για τη ζωή τους, να το και να μπορούν ως ανθρώπινα όντα να επωφεληθούν από όλες τις κατακτήσεις ε, των ε, ανθρώπων. Εκατό χρόνια βέβαια επέτειο σήμερα της Διεθνούς ε, Μέρας για την Γυναίκα. Πολλά έχουμε καταφέρει. Βρισκόμαστε εξάλλου σε μια περιοχή του κόσμου όπου πραγματικά υπήρξαν μεγάλες πρόοδοι και οι προσκεκλημένες μας ήδη το ανέφεραν Ωστόσο, ακόμα και έτσι, οι γυναίκες στην πολιτική ζωή λείπουν. Είμαστε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο 35% γυναίκες, ναι μεν, αλλά στα εθνικά μας κοινοβούλια, σε πολλά από τα εθνικά μας κοινοβούλια, πόρο απέχουμε από την επίτευξη τέτοιων στόχων. Και αυτό δεν αφορά μόνο την ε, κοινοβουλευτική πολιτική ζωή, αλλά και τις κυβερνήσεις, ε, τις τοπικές διοικήσεις, ε, όπου αυτό πραγματικά με παραξενεύει. Γιατί ενώ οι γυναίκες μπορούν να συμμετέχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση τόσο κοντά στα σπίτια τους, στη γη τους, γιατί δεν συμμετέχουν στην τοπική, στις τοπικούς μηχανισμούς. Θα πρέπει να προβληματιστούμε στις χώρες μας για αυτό το γεγονός και να δώσουμε κίνητρα για τη συμμετοχή των γυναικών στην τοπική πολιτική ζωή, στις περιοχές τους, στις περιφέρειές τους. Και με μια δεύτερη παρατήρηση ε, θέλω να επιστήσω την προσοχή γιατί βλέπουμε να υπάρχει κάποια οπισθοδρόμηση αυτή τη στιγμή. Η κρίση η οικονομική, η κοινωνική, η χρηματοπιστωτική έχει πάντα μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή των γυναικών. Βλέπουμε πως αυξάνεται η φτώχεια, η ανισότητα, οι διακρίσεις, οι δυσκολίες πρόσβασης των γυναικών στις θέσεις απασχόλησης με δικαιώματα αλλά και γίνονται και περικοπές στην κοινωνική πρόνοια, στις δημόσιες υπηρεσίες, στην παιδεία, στη στήριξη των οικογενειών, στη στήριξη των παιδιών, στη στήριξη των ηλικιωμένων. Και αυτό φυσικά έχει αντίκτυπο και πάλι στην συμμετοχή των γυναικών και στην πολιτική ζωή. Και ακριβώς σε τέτοιες επαιτίου, σε, τέ, σε τέτοιες ημερίδες θα πρέπει να το σημειώνουμε αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό να το θυμίζουμε στους πολιτικούς άνδρες και γυναίκες. Χρειάζεται αλληλεγγύη και θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τις πολιτικές αλλαγές ε, στη ζωή μας έτσι ώστε σε λίγα, σε λίγα χρόνια οι δικές μας διάδοχοι να μπορούν να πούν ότι αγωνιστήκαμε για την αλλαγή στην ζωή των γυναικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Φιγκερέντο. Ο η κυρία Τσαρούχα Κόλια είναι από το, από Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ε, θα ήθελα να, και εγώ να ενώσω τη φωνή μου και τους προβληματισμούς μου με ό,τι μέχρι τώρα έχει ακουστεί. Έχω συμμετάσχει πολλές φορές σε παρόμοιες ε, ε συνδιασκέψεις ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τιμάει που ακόμα και σήμερα ε, εκπροσωπώ τη χώρα μου μαζί με δύο άλλο, άλλους άξιους συναδέλφους ε, αγαπητές φίλοι, ε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, σε ό,τι αφορά τη χώρα μου, ε, ο έως τώρα αγώνας των γυναικών για την εξασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας σε σύγκριση με τους άντρες στη συμμετοχή στους τομείς άσκησης της πολιτικής αναγνωρίστηκε σε επίπεδο νομοθετικής εξουσίας και αποτυπώνεται σε μια σειρά σχετικών νομοθετημάτων. Αυτά παρτίζουν ένα ισχυρό ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αποτελεί ένα σταθερό πυλώνα και δημιουργεί μια κοινή συνισταμένη για την εξασφάλιση ουσιαστικής ισότητας σε θέματα εκπροσώπησης και άσκησης της πολιτικής, κυρίως μέσα από την καθιέρωση συγκεκριμένων ποσοστώσεων συμμετοχής των γυναικών σε όλους τους πολιτικούς τομείς της χώρας μου. Ε, ενδεικτικά αναφέρω ε, το νόμο ε, του 2000 που θεσπίστηκε για τη διασφάλιση της ισόρροπης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο δημόσιο στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ιδιωτικού δικαίου, όπως και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, ε, όπως επίσης και ένας νόμος ε, πρόσφατος του 2008 που καθορίζεται, όπου καθορίζεται ότι στους συνδυασμούς των κομμάτων ο ρυθμός των υποψηφίων από κάθε φύλλο οφείλει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 1 τρίτον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων βουλευτών στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας παρόλη όμως τη θέσπιση και την εφαρμογή των σχετικών νόμων και πολλών άλλων που δεν τους αναφέρω λόγω χρόνου η υφισταμένη κατάσταση αναφορικά με τη συμμετοχή των γυναικών στα πολιτικά κέντρα λήψης αποφάσεων αναδεικνύει μια μάλλον απογοητευτική εικόνα. Συγκεκριμένα στην παρούσα Βουλή, στην παρούσα σύνθεση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, μόνο 52 γυναίκες κατέχουν τη βουλευτική ιδιότητα σε σύνολο 300 βουλευτών σε ποσοστιαίο επίπεδο ο αριθμός αυτός μεταφράζεται στο 17,3% και είναι υψηλότερος που έχει σημειωθεί ως τώρα σε σύγκριση με τις εκλογές προηγούμενων ετών. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το ποσοστό των γυναικών ε, απέναντι στους άνδρες βουλευτές ανήλθε στο 16% το, 7, το 2007, στο 13% το 2004, στο 10% το 2002 και τέλος στις εκλογές του 1996 ήταν μόλις η συμμετοχή των γυναικών 6,3%. Στην Ευρωβουλή τα στοιχεία ε, είναι περισσότερο ενθαρρυντικά. Ε, συγκεκριμένα 7 γυναίκες κατέχουν ε, την ιδιότητα της Ευρωβουλευτού σε σύνολο 22 βουλευτών που εκπροσωπούν τη χώρα μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ποσοστό το οποίο έφτασε 31,8% σε σχέση με ευρωεκλογές του 9. Τώρα, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ε, στις πρόσφατες εκλογές ε, ε, του Νοεμβρίου του 2010 εξελέγησαν 32 γυναίκες μόνο δήμαρχοι σε σύνολο 1.033 δημάρχων όλης της χώρας. Ποσοστό δηλαδή 3,1% σε σχέση με τις δημοτικές εκλογές του 2006. Συμπτωματικά το ίδιο ποσοστό εκλογής γυναικών δημάρχων έχει καταγραφεί και στις πιο πρόσφατες εκλογές του 2010, συγγνώμη, αυτά που ανέφερα το, 3,1% είναι το 2006. Το 2010, τις πρώτες εκλογές, εξελέγησαν 9 συνολικά γυναίκες, σε, συνολικό, σε γενικό σύνολο 325 δημάρχων, ε, μηδενικά ποσοστά υποψηφίων γυναικών περιφερειαρχών, καταγράφηκαν στις ίδιες εκλογές, σε συνολικό ρυθμό 13 δηλαδή, δεν υπάρχει καμία γυναίκα εκλεγμένη περιφερειάρχης, ενώ εξελέγησαν 11 γυναίκες αντιπεριφερειάρχες, σε σύνολο 57 αριθμός μεταφράζει ποσοστό της τάξης του 19,3. Ε, Όλα τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός ζητήματος με διακριτές κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις στη χώρα μου και αποδεικνύουν την ανάγκη αύξησης των προσπαθειών εκείνων οι οποίες οφείλουν να στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στη διεκδίκηση πολιτικής εξουσίας στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο όμως θα πρέπει αδιάρρηκτα να συνδυαστεί με τη βελτίωση του εχώριου κλίματος και συγκεκριμένα την ενθάρρυνση, όπως ήδη είπατε κι εσείς αγαπητές φίλες, ε, την ενθάρρυνση του συνόλου των Ελλήνων ψηφοφόρων προς την κατεύθυνση στήριξης ερετών γυναικών σε δημοτικό, περιφερειακό και γενικότερα σε εθνικό επίπεδο. Χωρίς να θέλω ε, να, υποτιμήσω το σύνολο των αλλαγών που έχουν επιτευχθεί κυρίως σε νομοθετικό επίπεδο, δεν μπορώ παρά να σημειώσω ότι η ισότητα των γυναικών στο κρίσιμο αυτό πεδίο έχει κατακτηθεί περισσότερο τυπικά παρά ουσιαστικά και πέρα από την αδιαφυσβήτητη επιτυχία της αύξησης της συμμετοχής των γυναικών σε σημαντικούς τομείς της σύγχρονης κοινωνικής ζωής στην Ελλάδα, όπως την εκπαίδευση στην εργασία, ένα σύνολο παραγόντων όπως οι υφιστάμενες συντηρητικές προκαταλήψεις, γενικότερα συμφέροντα, αλλά και επίσης η παθητική στάση των γυναικών σχετικά με την ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά εμποδίζει την περαιτέρω πρόοδο και εξέλιξη αναφορικά με το θέμα της σημερινής διακοινοβουλευτικής μας συνάντησης. Ε, θα μπορούσα να συμπληρώσω πολλά και πολλούς προβληματισμούς που ήδη ακούστηκαν. Η, κρίση οικονομική που διέρχεται και η χώρα μου σε αυτή την δύσκολη ε, συγκυρία ε, πρώτο ε, που χτυπάει είναι τη γυναίκα. Οι περισσότερες άνεργες ε, στη χώρα μου από τους ανέργους είναι γυναίκες και νέες γυναίκες και γυναίκες επιστήμονες. Έτσι, μέσα από τις παρούσες συνθήκες οι όποιες λύσεις αποφασιστούν να δρομολογηθούν θα επιτύχουν εάν έχουν τη βάση τους στη λογική ενός ισορροπημένου κοινωνικού μοντέλου το οποίο θα προτάσει και το ηθικό δικαίωμα της απρόσκοπτης και ουσιαστικής εφαρμογής της αρχής της ισότητας των δύο φύλων σε όλες τις εκφάνσεις της σύγχρονης κοινωνικής ζωής της χώρας μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Μουρέν Σαπιές, η οποία είναι μέλος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επίσης αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Γυναικών. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Merci, Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που διοργανώσατε αυτήν την ε, ημερίδα και ευχαριστώ τις δύο προέδρους που ήρθαν ε, στο έδρανο ε, και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο για να αντιπροσωπεύσουν τον αγώνα υπέρ των γυναικών. Το πρώτο σημείο για το οποίο θα ήθελα να παρέμβω, κυρία Πρόεδρε, είναι να υπογραμμίσω ότι πρόκειται για ένα συλλογικό αγώνα, ένα κοινωνικό αγώνα, έναν αγώνα των καιρών μας. Δεν πρόκειται για έναν αγώνα της αριστεράς ή της δεξιάς δεν είναι ένας αγώνας ανδρών ή γυναικών, είναι ένας αγώνας τον οποίο πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί. Ποια κοινωνία θα μπορούσε να στερηθεί σήμερα το 50% της ενεργειάς της, 50% της ευφυΐας της και ωστόσο σήμερα αυτό είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Και αυτό είναι μια πρώτη παρατήρηση που θα πρέπει να την συνειδητοποιήσουμε γιατί είναι αυτό ζήτημα που αποσχολεί όλους μας. Ε, και κοιτάξτε, πόσο τα κράτη, οι οικογένειες κάνουν προσπάθειες για την κατάρτιση των κοριτσιών, για την ισότιμη κατάρτιση των ανδρών και των ε, γυναικών, των αγοριών μάλλον και των κοριτσιών τους. Και λίγα χρόνια αργότερα, μετά από λίγα χρόνια στα διαδρομίας, δείτε πόσο αποκλίνει η... Ε, η εξέλιξή τους. Πόσο δηλαδή διαφορετική είναι η εξέλιξη των παιδιών αυτών για τα οποία όλοι προσπαθήσαμε. Και αυτό το λέω ενώπιον των συναδέλφων ε, το, της Επιτροπής Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Δεν υπάρχουν ε, σύνορα. Όλοι μαζί σε αυτό την Επιτροπή κάνουμε αυτόν τον αγώνα προς την ίδια κατεύθυνση. Σίγουρα δεν προχωράμε αρκετά γρήγορα. Έχετε δίκιο, κυρία Πρόεδρε. Θα θέλαμε αυτή η Επιτροπή να μην είναι μια Επιτροπή κατά κάποιο τρόπο ουδέτερη, προσαρτημένη, δευτερεύουσα. Θα έπρεπε να είναι μια Επιτροπή η οποία θα γίνεται σεβαστή από όλε τι άλλε και ίσω κάποια ημέρα των ημερών να μην χρειαζόμαστε πια αυτή την Επιτροπή. Δεύτερη παρατήρηση που ήθελα να κάνω είναι ότι πολύ θα ήθελα γυναίκες ε, μέσω των δεξιοτήτων τους και των ικανοτήτων τους να φτάσουν σε μια θέση απόλυτα ίση με αυτή των ανδρών στην κοινωνία μας. Είναι το όνειρό μου και θα πρέπει να πω ότι κάποιες στιγμές αμφισβήτησα την πολιτική, τη, μάλλον είχα αμφιβολίες για την πολιτική των ποσοστώσεων, γιατί θεωρούσα πως ήταν κάπως μειωτικό για μια γυναίκα να χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τις ποσοστώσεις ε, για να φτάσει σε κάποια θέση. Αλλά σήμερα λέω ότι δεν θα τα καταφέρουμε χωρίς τις ποσοστώσεις και γι' αυτό και εκτιμώ αυτό που είπε ο Πρόεδρος Μπούσεκ πριν από λίγο, που είπε δηλαδή ότι η Ευρώπη θα πρέπει να πατήσει κάπως τον γκάζι για να οθήσει τα κράτη-μέλη προς αυτήν την κατεύθυνση. Και όπως είπε και η Ελληνίδα συνάδελφος πριν από λίγο, για να μπορέσουν έτσι οι γυναίκες να προχωρήσουν σε αυτή την κοινωνία όπου πρέπει να έχουν μια ισότιμη θέση με τους άνδρες. Και ανησυχώ. Ανησυχώ. Και η Νικόλ Φοντέν το είπε πριν από λίγο. Γιατί τα πολιτικά κόμματα προτιμούν να πληρώνουν τα ισχυρώσει του ε, παρά να αφήσουν το χώρο στι γυναίκε. Μα τι φοβούνται την ε, ανταγωνισμό των γυναικών. Φοβούνται τη δέσμευσή του, την προσήλωσή του, την αίσθηση τη εργασία, την εργατικότητά του. Γιατί να φοβούνται. Πρέπει όλοι μαζί να προχωρήσουμε ήρεμα και αποτελεσματικά. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το μέλλον όλων μας ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη εξαρτάται από την δύναμη πυθούς. Και Ανησυχώ όταν βλέπω κάποιες περιφερειακές μεταρρυθμίσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη την θέση που πρέπει να δοθεί στις γυναίκες σε αυτές τις ε, μελλοντικές μεταρρυθμίσεις. Η τρίτη παρατηρήση επί της οποίας θέλω να παρέμβω είναι αυτό που προέκυψε πριν από κάποιες μέρες μια έρευνα που έλεγε ότι παντού οι άνδρες πιστεύουν ότι, μάλλον το 20% των ανδρών πιστεύει ότι σε περίπτωση κρίσης η προτίμηση στην απασχόληση, για μια θέση μάλλον απασχόληση, θα πρέπει να δοθεί στους άνδρες. Τέτοιου είδους έρευνες ε, θα μας δείχνουν ότι <laughs> έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας για να καταστεί, για να κάνουμε χώρο για τις γυναίκες όχι μόνο στην πολιτική αλλά και στον, χώ... στον κόσμο της εργασίας. Μιλάμε σήμερα για τη θέση της γυναίκας στην πολιτική, αλλά θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου και ότι θα πρέπει μετά από αυτό να μιλήσουμε και για την θέση της γυναίκας στον κόσμο της εργασίας για να μην την μεταχειρίζονται διακριτικά στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία. Τέλος, θα ήθελα να σας πω ακόμα κάτι. Πόσο καιρό ακόμα θα φεθούμε και θα δεχόμαστε οι γυναίκες να έχουν τόσο χαμηλότερου μισθού από τους άνδρες. Το βρίσκετε εσεί φυσιολογικό, κύριοι και κυρίες, κυρίες και κύριοι, στην κοινωνία μας να χρειάζεται πέντε χρόνια μια γυναίκα για να κερδίσει το, το μισθό που κερδίζει ένας άντρας σε τέσσερα. Εγώ όχι, δεν το βρίσκω φυσιολογικό και πραγματικά θα, ντρα, θα ντρεπόμουν να αφήσω αυτή την κληρονομιά στα εγγόνια μου που είναι και μάλιστα πολλά. Και πιστεύω πως έχουμε πολλή δουλειά, Πρόεδρε, μπροστά μας. Θα ήθελα να σας προτείνω μετά από τις εργασίες σε κάποια κράτη και σκέφτομαι κυρίως αυτό που έκανε η Ζιζέλα Λιμή να μπορέσουμε να δουλέψουμε για τη ρήτρα της πιο ευνοούμενης Ευρωπαίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Χιμενές έχει το λόγο τώρα. Sí. Eh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ως ε, γυναίκα βουλευτής και μέλος της Επιτροπής των Πολιτικών Ελευθεριών χαίρομαι που μπορώ να εορτάσω αυτή την ημέρα με διακεκριμένες προσωπικότητες των γυναικών. Είναι αναπόφευκτο ε, να συλλογιστούμε τις, ε, τα ορόσημα στην ιστορία του γυναικείου κινήματος όπως στη Νέα Υόρκη όπου χιλιάδες γυναίκες ε, διατύπωσαν ε, θεμελιώδη δικαιώματα. Οι σουφραζέτες μπορεί να αποτελούν ιστορία σήμερα, αλλά παρόλα αυτά αντιμετωπίζουμε πολλά από τα αιτήματά τους ακόμα. Ε, το θέμα της ε, μικρότερης αμοιβή. Το θέμα του συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής είναι ένα τεράστιο μέτωπο όταν μιλάμε για ισότητα. Έχουμε δικαίωμα ψήφου πλέον, αλλά η πολιτική συμμετοχή των γυναικών, όπως είπαν πολλοί ήδη, εξακολουθεί να είναι περιορισμένη και ακόμα έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε. Δεν θέλουμε να μας χαρίσουν τίποτε, ούτε όμως θα επιτρέψουμε να μας αρνούνται πράγματα που δικαιούμεθα. Λόγω προκατάληψης, λόγω άγνοιας, λόγω φόβου ότι δεν θα μπορούν να συνδυάσουν ζωή και, ε, επαγγελματική ζωή και οικογένεια οι γυναίκες. Βεβαίως ξέρουμε το τίμημα που πρέπει να πληρώνουμε και ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι ε, που εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο που θεωρούνται υποδέστερες. Θέλω να καταγγείλω δημοσία την ε, αντιμετώπιση πολλών γυναικών στις Ισλαμικές χώρες όπου οι διακρίσεις κατά των γυναικών είναι μια πραγματικότητα δύσκολο να γίνει κατανοητή. Εξανίσταμε κατά της, ε, των διακρίσεων στις αραβικές χώρες Πώς είναι δυνατόν να καταλάβει κανείς ε, της, ε, την αντιμετώπιση των γυναικών που λιθοβολούνται λόγω ή που ε, τους ρίχνουν οξύ στο πρόσωπο ή τις αντιμετωπίζουν στα πλαίσια βομβιστικών ενεργειών. Ε, θα πρέπει αυτό να αντιμετωπιστεί και στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό να δούμε το ρόλο που πρέπει εμείς να παίξουμε στην προστασία των νέων γυναικών που ζουν στην Ευρώπη και θέλουν να ε, ακολουθήσουν το δικό μας πρότυπο ζωής ενώ δεν τους επιτρέπεται γιατί πολλοί Άραβες ή Μουσουλμάνοι θέλουν να παραμείνουν περιθωριοποιημένοι στις ευρωπαϊκές πόλεις. Χρειάζονται χρόνια για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα. Ανησυχώ επίσης πολύ με το θέμα της βίας στο σπίτι κατά των γυναικών. Τα θύματα αναφέρθηκε σήμερα δεν αντιμετωπίζονται με την προτεραιότητα που χρειάζονται από το Κοινοβούλιο μας. Πρέπει να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη προστασία και ελπίζω να ψηφίσουμε σχετικά μέτρα. Πρέπει να προασπίσουμε τα δικαιώματα των γυναικών, ε, διότι αυτό έχει σχέση με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ε, Ενωμένη Ευρώπη με κοινέ αξίες μεταξύ ανδρών και γυναικών όλοι θα πρέπει να έχουν δικαίωμα στην ελευθερία και στην ε, αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ. Κυρία Πλάμ. Το λόγο στην κυρία Πλάμ η οποία είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές και τις ομιλήτριες για τα μηνύματά τους. Πάνω απ' όλα όμως θέλω να ευχηθώ καλή επέτειο, ευτυχισμένη 8η Μαρτίου για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια στον κόσμο. Γνωρίζουμε όλοι ότι πέρασαν ήδη 100 χρόνια. 100 χρόνια προσπαθειών, αγώνων, πρόοδου, Όλοι συμμετείχαμε στους αγώνες και όλοι μοιραστήκαμε τις επιτυχίες, τις προόδους αλλά και τις αποτυχίες. Γυναίκες και άνδρες συνέβαλαν. Δεν νομίζω ότι η ισότητα των φύλων είναι μόνο θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης είναι περισσότερο ένα εργαλείο, ένα μέσον για αποτελεσματικότητα και πρόοδο. Είναι ένας τρόπος επιτέλους να επιτύχουμε την Ενωμένη Ευρώπη. Μια Ευρώπη με ευθυδικία, δικαιοσύνη για όλους τους πολίτες. Άκουσα με μεγάλη προσοχή συναδέλφους που μίλησαν για τις αρνητικές επιδράσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης στις γυναίκες Πράγματι, η φτώχεια ε, πλήττει περισσότερο τις γυναίκες, όπως και η μετανάστευση. Οι διακρίσεις στην αγορά εργασίας βαθαίνουν, οι διακρίσεις στην κοινωνία επίσης. Και αν θέλουμε πράγματι η Ευρώπη να πατήσει γκάζι, όπως είπατε, όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να στείλουμε ισχυρό μήνυμα. Το 2009 ε, τέθησε ισχύ η νέα συνθήκη της Λισαβόνας. Σύμφωνα με τη συνθήκη αυτή έχουμε το δικαίωμα να αναλάβουμε νομοθετικές πρωτοβουλίες και μιλώ για, και για πρωτοβουλίες πολιτών εδώ. 27 κράτη-μέλη μπορούν. Ας οργανώσουμε εκστρατείες παντού στην Ευρώπη. Ας φέρουμε τις γυναίκες πιο κοντά σε μας. Η κυρία Νικόλ Φοντέν μίλησε για την αλληλεγγύη. Πολύ σημαντική είναι η αλληλεγγύη εδώ. Θα πρέπει να συνενώσουμε όσο γίνεται περισσότερους άνδρες και γυναίκες. Ας οργανώσουμε τέτοιες εκστρατείες, ας συλλέξουμε υπογραφές, ας ε, επιβάλλουμε τις ποσοστάωσεις. Γιατί, κυρία Ρόμπινσον, δεν πιστεύω ότι υπάρχει πλήρη συνείδηση σε όλη την Ευρώπη τη σημασία της γυναικείας συμμετοχής στα πολιτικά. Το 90% των Γάλλων σήμερα πιστεύουν ότι η παρουσία των γυναικών στην πολιτική είναι πολύ σημαντική. Δεν αρκεί αυτό. Ας δείξουμε ότι οι στατιστικές όντως είναι πραγματικότητα. Ας αρχίσουμε να μαζεύουμε υπογραφές και μέσα από πρωτοβουλία πολιτών ας εφαρμόσουμε, ας εισαγάγουμε και ας επιβάλλουμε τις ποσοστώσεις. Γιατί το άλλο μισό της κοινωνίας, εμείς δηλαδή οι γυναίκες, θα πρέπει να εκπροσωπείται στην πολιτική. Δεν θέλουμε να μπούμε στην πολιτική μόνο για τα αξιώματα και τις υψηλόβαθμες θέσεις θέλουμε γιατί θεωρούμε ότι έχουμε καλύτερες απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας και τα προβλήματα των γυναικών στην κοινωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γκόμες, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ κυρία Γκόμες, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. θα ήθελα να χαιρετήσω τις ε, εισηγήτριες και όλο ιδιαίτερος ε, την Νικόλ Φοντέν και τη μέρη Ρόμπινσον που θα μπορούσε να είναι και υποψήφια, όπως γνωρίζουμε, για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έγινε το 2009, αλλά μπορεί και ελπίζω να γίνει στο μέλλον, γιατί χρειαζόμαστε γυναίκες γυναίκες σε θέσεις ε, ορατές, σε θέσεις ε, λήψης αποφάσεων για να υπάρξει διαφορά, να μπορέσουν να σημάνουν τη διαφορά για μια ατζέντα ε, που θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των γυναικών. Πιο συγκεκριμένα, η κρίση οικονομική την οποία ζούμε στην Ευρώπη και η οποία είναι ιδιαίτερα σοβαρή σε μερικές χώρες όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, μας κάνει να δούμε πως οι γυναίκες είναι πραγματικά οι πρώτες που υποφέρουν από τις συνέπειες. Είναι αυτές που θυσιάζονται, χάνουν τη δουλειά τους, πέρα από τη διαφορά των μισθών που ούτως ή άλλως υπήρχε, αλλά εδώ υπάρχει μια ευκαιρία. Υπάρχει μια ευκαιρία να δούμε ποιο είναι ο ρόλο που μπορούν να παίξουν οι γυναίκε στα όργανα λήψη οικονομικών αποφάσεων, στα μεγάλε τράπεζε και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μα, Δηλαδή, όχι μόνο στην εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική ζωή, που είναι πράγμα πολύ, πολύ σημαντικό φυσικά, αλλά θα πρέπει να δούμε ε, πώ θα μπορέσουν να εκπροσωπηθούν και στα όργανα που έχουν ε, οικονομική εξουσία και που κατά συνέπεια έχουν και πολιτική επιρροή. Ε, να μπορέσουμε δηλαδή να σχηματίσουμε στρατηγικές και να τις ασκήσουμε ώστε να υπάρξουν περισσότερες γυναίκες και σε αυτούς τους οργανισμούς και να παίξουν καθοριστικό ρόλο για ε, τα θέματα αυτά που επηρεάζουν τόσο πολύ την κοινωνία. Ε, παραδόξως Πολλοί κόσμος ε, στο... Ε, στην οικονομία πιστεύει πως αν υπήρχαν περισσότερες γυναίκες ε, στις τράπεζες δεν θα είχαν οδηγηθεί σε τέτοια άκρα, σε πράγματα δηλαδή τόσο καταστροφικά. Πιστεύω επίσης πως είναι πολύ σημαντικό για μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για το Ευρωκοινοβούλιο γιατί έχουμε την Επιτροπή Ισότητας που είναι ένα σημαντικότατο βήμα εμπειρογνωμοσύνης και επαγρύπνησης για τα θέματα που αφορούν την προώθηση της ισότητας για τις γυναίκες αλλά θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική ώστε να τοποθετήσουμε γυναίκες εκεί όπου μπορούν να έχουν επιρροή μέσω της δικής τους ευαισθησίας και μέσω της δικής μας ε, βοήθειας. Ε, και βεβαίω ένα άλλο τομέα πολύ σημαντικό είναι, ένας είναι ο τομέα τη ε, ασφάλεια και, και της άμυνας είναι ένας τομέας όπου συνήθω και παραδοσιακά οι άντρες καθορίζουν τα όσα συμβαίνουν όμως είναι ένας τομέας που έχει μεγάλες επιπτώσεις για την κοινωνία μας και για την οικονομία μας χρειαζόμαστε δηλαδή περισσότερες γυναίκες επιρογνώμονες σε αυτούς τους τομείς όχι μόνο γιατί αυτό έχει επίπτωση στην οικονομία αλλά γιατί σε τελική ανάλυση είναι σημαντικοί ε, παράγοντες στα θέματα πολέμου και ειρήνης Τέλος, να πω επίσης ότι σε μια νέα πολιτική που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει τους γείτονές της αλλά και ολόκληρο τον κόσμο θα πρέπει να αποκομίσει διδάγματα από τις ασυνέπειες, τις υποκρισίες, τις την, την ε, ασυνέπεια που βλέπουμε και που διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή στην Βόρεια Αφρική γιατί η πολιτική γυτνίαση πέρα από τα ωραία λόγια για πρόθεση της δημοκρατίας, για ισότητα, για ανθρώπινα δικαιώματα κτλ στην πράξη δεν κατάφερε και πολλά από αυτά τα πράγματα, αλλά στην ουσία υποστήριξε δικτατορίες, δικτατορικά καθεστώτα. Θα έπρεπε λοιπόν με αποφασιστική συμμετοχή των γυναικών να απαιτήσουμε τη δημοκρατία, δικαιώματα και ελευθερίες. Γυναίκες στον αραβικό κόσμο, στον ισλαμικό κόσμο που θα αποδείξουν ότι το Ισλάμ δεν είναι ασύμβατο με τις δημοκρατικές πεπιθήσεις θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά, ε, σε όλα αυτά να συμμετέχουν οι γυναίκες και να επηρεάσουν και τις ευρωπαϊκές πολιτικές ε, γυτνίασης με αυτές τις χώρες και να ενθαρρύνουν τη διαδικασία της δημοκρατικής μετάβασης η οποία δεν θα υπάρξει εάν δεν υπάρξουν ε, δεν υπάρξει συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ η κυρία Κολάκα Βομπίνσκα, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ. Δεν έχουμε τίποτα. Ε, ε, ε, κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, καλά διαγνώσαμε το πρόβλημα. Ξέρουμε που εντοπίζονται οι ανισότητες, ξέρουμε το πρόβλημα των αμοιβών, αλλά το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξει όσο γίνεται ταχύτερα η κατάσταση. Να πω το εξή. Αν οι γυναίκες μόνες τους ε, δεν παλέψουν, ε, δηλαδή ενώ οι ίδιες αν δεν παλέψουν για την αλλαγή της νομοθεσίας, δεν θα πετύχουμε και πολλά πράγματα. Πριν από τρία χρόνια στην Πολωνία ε, δημιουργήσαμε ένα συνέδριο γυναικών και χάρη στη δουλειά αυτή τη τριετούς περίοδου καταφέραμε κάποια, να ισχύσουν κάποιες ποσοστώσεις σε όλες τις επόμενες εκλογές. Συναντήσαμε μεγάλη αντίσταση, άρα άρχισε μια μεγάλη συζήτηση σε όλη τη χώρα, γιατί η μάχη για την ισότητα δεν είναι μόνο για τη θέση των γυναικών στην πολιτική, αλλά αγώνας για αλλαγή νοοτροπίας στην κοινωνία γενικότερα. Αυτή λοιπόν η αντιπαράθεση συζήτηση άλλαξε άρδιν τον τρόπο σκέψης της κοινωνίας μας και τον τρόπο σκέψης κάποιων πολιτικών. Ε, καταφέραμε να αλλάξουν πολλά και νομοθετικά. Δεν τα καταφέραμε όλα γιατί θέλαμε 50% ισότητα 50-50 δηλαδή. Είμαστε τώρα στο 35% και φέτος θα γίνουν βουλευτικές εκλογές σύμφωνα με τον νέο εκλογικό νόμο. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Πού να τις βρούμε τις γυναίκες υποψήφιες ε, ε, βουλευτίνες. Γυναίκες που δεν θα ε, φοβούνται, που θα έχουν αυτοπεποίθηση, που θα νιώθουν ότι έχουν αρκετές ικανότητες για να αναλάβουν αυτή την υποχρέωση. Είναι και αυτό. Θέλω όμως να σας καλέσω το Σεπτέμβριο στην Πολωνία για ένα δεύτερο συνέδριο των γυναικών. Θα είναι διεθνής διάσκεψη αυτή τη φορά γιατί αναλαμβάνει η Πολωνία την Προεδρία της Ένωσης και θέλουμε να καταλήξουμε σε νέους στόχους, γιατί είμαστε ένα μαζικό, αυθόρμητο εν πολύ κίνημα, δεν είμαστε δηλαδή οργάνωση κανονική, είμαστε ένα μαζικό κίνημα και θέλουμε να συμφωνήσουμε σε στόχους που θα προωθήσουμε στις μετέπειτα πολιτικές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις και ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί πολλά να κάνει διότι μπορεί να υποβάλει προτάσεις, νομοθετικές πρωτοβουλίες, εκθέσεις, αποφάσεις. Αν δεν υποστηριχθούν τέτοια μαζικά κινήματα στα κράτη-μέλη μας, δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Τάγμα Σούμάχερ θα πάρει το, το λόγο. Παρακαλώ, έχετε. Thank you very much, um, Chair. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να κάνω τέσσερις παρατηρήσεις. Πρώτον, να συγχαρώ όλες τις γυναίκες και τους άνδρες στον κόσμο για την δέσμευση τους υπέρ της ενίσχυσης των γυναικών. Να συγχαρώ και την Επιτροπή Γυναικών για την σημερινή εκδήλωση. Η παραμέληση των ε, δικαιωμάτων των γυναικών σημαίνει ότι υποαξιοποιείται το μισό πληθυσμιακό δυναμικό και στην επιστήμη και στην τεχνολογία και στο εμπόριο και στις ε, νευτικές διαπραγματεύσεις και παντού θα πρέπει να αξιοποιηθούν σε όλο τον κόσμο. Ελάχιστες γυναίκες συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για την ειρήνη, για την αλλαγή του κλίματος, για το εμπόριο. Μία εστίαση των γυναικών θα είναι η διεύρυνση της συμμετοχής των γυναικών. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε για να κλείσει το κενό στη συμμετοχή γυναικών σε ένα σωρό τομείς και να αξιοποιήσουμε τα ωφέλη από τη συμμετοχή για την κοινωνία γενικότερα. Και προσβλέπουμε στην συνεχιζόμενη στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γι' αυτό σε θέματα όπως να σταματήσει η βία κατά των γυναικών που και άνδρες και γυναίκες θα πρέπει να στηρίξουν στεναρά. Η επικείμενη επίσκεψη της Μισελ Μπασιλέ στι Βρυξέλλες θα ενισχύσει τη συνεργασία σε αυτό το τομέα. Θέλω να αναφερθώ και σε μια ιστοσελίδα την, το Διεθνές Δίκτυο Γυναικών στην Πολιτική για τη Γνώση. Είναι ένα επιγραμμικό ε, πρόγραμμα, μια πλατφόρμα ε, με πρόσβαση σε όλους στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για να προωθηθούν οι γυναίκες στην πολιτική ζωή. Τελευταίο θέμα που θέλω να αναφέρω, συνεχίζοντας αυτά που ακούσαμε σήμερα το πρωί και που έχει σχέση με την Βόρεια Αφρική, εδώ οι γυναίκες βλέπουν παράθυρο ευκαιρίας για να αποκτήσουν περισσότερο η εξουσία πολιτική οι γυναίκες γιατί ανοίγονται τώρα οδοί για μεταρρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τη συμμετοχή των γυναικών ε, ε, στην περιοχή θα ενισχυθεί δηλαδή η αίσθηση και η ιδιότητα του πολίτη μεταξύ των γυναικών στον αραβικό κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Εκπρόσωπος τώρα του European Women Lobby θα πάρει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εδώ και χρόνια αγωνιζόμαστε για τις γυναίκες σε όλη την Ευρώπη και δι για την ισότητα. Μιλήσαμε πολύ για την ποσόστοση σήμερα το πρωί. Η ερώτηση είναι η εξή. Θα ήταν ε, δυνατό, εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή κάποιοι περιορισμοί. Ε, θα ήταν δηλαδή νομικά και πολιτικά δυνατό. Επίσης αναφέρει και το θέμα της αλληλεγγύης, ο αγώνας από κοινού μήπως θα μπορούσε ένας αγώνας από κοινού με άνδρες και γυναίκες θα μπορούσε να γίνει και εδώ πέρα, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τις επόμενες ευρωεκλογέ. Θα επιθύσαμε να γίνει κάτι τέτοιο, μια συμμαχία σε όλα τα πολιτικά κόμμα και με την υποστήριξη φυσικά της κοινωνία των πολιτών και της οργανώσει των γυναικών, ούτω ώστε να επιτευχθεί ισότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις επόμενες εκλογέ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα να πω το εξής, ότι καταρχήν ευχαριστώ τις καλεσμένες μας, ευχαριστώ όλους όλες όσοι συμμετείχαν σε αυτήν εδώ τη συζήτηση, ε, ενδιαφέρουσες απόψεις ακούσαμε και τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της ε, συνεδρίασής μας. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ τους καλεσμένους μας. Τώρα το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με το εξή. Εμείς θα ανταλλάξουμε εμπειρίες, να δούμε δηλαδή πώς ο καθένας δουλεύει στη χώρα του, ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές για τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική. Και εκ των προτέρων να ευχαριστήσω ε, όλα τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων που έχουν περιγράψει τις δικές τους εμπειρίες και τα οποία μέλη είναι έτοιμα, διαθέσιμα να μας ενημερώσουν για αυτή την εμπειρία. Εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα να είχαμε τη συμμετοχή όλων στο πάνελ, αυτό ενημερωτικά, αλλά να πω το εξή. Όλοι, όλες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν το λόγο μετά από την εισαγωγή που θα γίνει και με αυτόν τον τρόπο να ενημερώσουν για την δική τους εμπειρία. Τώρα, να καλωσορίσω τον επόμενο ομιλητή, ή μάλλον ομιλήτρια, την κυρία Νέλε Λίνεν, που ήταν πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής για Ισότητα ε, Ευκαιριών Άνδρες-Γυναίκες, από την, τη Γερουσία, στο Βέλιο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και λίγοι κύριοι που είστε εδώ, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τον πολιτικό ρόλο των γυναικών στη Μελλοντική Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ακόμα αναγκαίο να διαφοροποιούμε μεταξύ ανδρών και γυναικών όταν μιλάμε για πολιτική δεν είμαστε πια ήδη ε, ισχυρές, ανεξάρτητες Ευρωπαίες γυναίκες. Είμαστε βεβαίως, αλλά το έργο μας ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Γι' αυτό και αυτές οι συναντήσεις παραμένουν πολύ σημαντικές για να εμπλουτίζουν τη γνώση μας για τη θέση των γυναικών και στην πολιτική και στην κοινωνία. Ο αριθμός των γυναικών πολιτικών μπορεί να αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, αλλά ακόμα μένουν πολλές προκλήσεις. Είναι γνωστό ότι οι γυναίκες λιγότερο αυθόρμητα δέχονται προαγωγές και ανώτερες και ανώτετες θέσεις. Το ίδιο και για την πολιτική εντολή. Οι γυναίκες στους εκλογικούς καταλόγους, στα ψηφοδέλτια θα πρέπει να, να μην θεωρούνται αναγκαίο κακό, αλλά ένα πλεονέκτημα. Ε, όταν εργάζονται μαζί άνδρες και γυναίκες βελτιώνουν τις επιδόσεις τους. Ε, η δημοκρατική κοινωνία επίσης προποθέτει ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους του τομεί και στι πολιτικές αποφάσεις. Οι σκανδιναβικές, οι βόρειες χώρες γενικά έχουν καλύτερη εκπροσώπηση, πιο ισότιμη και πιο ισορροπημένη κοινωνία. Πιστεύω λοιπόν ότι η καινοτομία και η δημιουργικότητα ε, ανεβρίσκονται εκεί όπου συνεργάζονται άνθρωποι με διαφορετικό υπόβαθρο. Ε, ως πρόεδρος της Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών στην Βελγική Γερουσία, ε, ένα βασικό θέμα είναι ίσες ευκαιρίες. ξέρετε ότι οι γυναίκες ε, με ε, επιχειρηματική κουλτούρα γυναικεία ε, είναι πιο δυναμικές, ανταγωνιστικές και καινοτόμες από ότι οι επιχειρήσεις με ανδρική επιχειρηματική κουλτούρα. Αυτό δεν είναι σλόγγαν από κάποιο λόμπι γυναικών, φεμινιστριών, αλλά προέρχεται από τα συμπεράσματα έκθεσης, η οποία ε, κατατάσσει και βαθμολογεί τις χώρες σε σχέση με το κενό ε, μεταξύ των φύλων. Ε, περισσότερες ε, ε, γυναίκες ε, από ό,τι δείχνει δέχονται την ε, μερική απασχόληση. Όχι από ελεύθερη επιλογή, αφού η, περισσότερη, η λιγότερη δουλειά σημαίνει λιγότερο εισόδημα, λιγότερη σύνταξη. Ε, κανείς δεν το επιλέγει αυτό με ελεύθερη επιλογή, αλλά κατά ανάγκη. Έτσι λοιπόν, ως πρόεδρος της Βελγικής Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών, ζητώ από τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη να βοηθήσουν την προσπάθεια για ίσες ευκαιρίες, να συμμετάσχουν στον αγώνα κατά των διακρίσεων στις αμοιβέ, να επιμείνουν οι τομείς με σοβαρή υποεκπροσώπηση γυναικών σε ηγετικές θέσεις, να ε, να, ενισχυθεί. Ε, αυτή είναι η, η άποψή μου, αλλά είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω εσείς τι πιστεύετε και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε την κυρία Λέινεν. Ε, επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Αλένα Γκαϊτζούσκοβα, αντιπρόεδρος η κυρία της Γερουσίας στη Τσεχία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Hezký den, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Mě je skutečně velkou ctí zúčastnit se tady tohoto Κυρία Πρόεδρε, αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μεγάλη τιμή συμμετοχή σε αυτήν την συνεδρίαση με αφορμή την εκατοστή επέτειο του αγώνα των γυναικών για ισότητα ευκαιριών και τα ίσα δικαιώματα. Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι βρίσκομαι δίπλα σε συναδέλφους όπως η Μαρλένε Ρούπρεχτ από την, με, με την εκπρόσωπο των γυναικών στο Συμβουλίο της Ευρώπης και άλλους συναδέλφους. Χαίρομαι πολύ που μπορώ και εγώ να συμβάλλω στη συζήτηση και μπορώ να παρουσιάσω μέρος της εμπειρίας μου από την Τσεχία. Ε, εμείς στην Τσεχική Δημοκρατία είμαστε περήφανες ως γυναίκες γιατί από τις πρώτες αποκτήσαμε το δικαίωμα ψήφου το οποίο δόθηκε το 1920 στις γυναίκες ε, το δικαίωμα να, εκλέγουν, να ψηφίζουν οι γυναίκες. Όμως από τότε και μετά δεν επιτελέσαμε και πολύ μεγάλη πρόοδο όσοι θα θέλαμε. Στην Τσεχία πέρσι ε, είχαμε το super, τη σούπερ εκλογική χρονιά το 2010 της, ε, το, την ήταν οι βουλευτικές μετά το φθινόπωρο για οι εκλογές, οι αυτοδιοικητικές και για τη γερουσία. Τα εκλογικά αποτελέσματα από τις τρεις αυτές εκλογές και ιδιαίτερα η σύνθεση των ψηφοδελτίων επιβεβαίωσαν και πάλι ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα θετικά αν θετικών διακρίσεων, δηλαδή για την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στην πολιτική. Αυτά τα μέτρα είτε τα κόμματα τα ίδια θα τα λάβουν ή θα τα συμπεριλάβει ο εκλογικό νόμος. Το πολιτικό σύστημα σήμερα δεν υποστηρίζει καθόλου, δεν προωθεί καθόλου τις γυναίκες. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τα ψηφοδέλτια, όπου βλέπουμε γυναικεία ονόματα, αλλά τα κόμματα τα δικούν άνδρες και στα ψηφοδέλτια ε, ε, βρίσκονται γυναίκες, ε, όχι όμως σε εκλόγιμες θέσεις. Οπότε, αν κάποιος θέλει να ψηφίσει μία γυναίκα, θα πρέπει να δώσει προτιμησιακή ψήφο. Στις τελευταίες εκλογές στην Τσεχία οι προτιμησιακές ψήφοι ελήφθησαν περισσότερο υπόψη και γι' αυτό ο αριθμός των γυναικών στο Κοινοβούλιο αυξήθηκε. Τώρα έχουμε επιτύχει αριθμό ρεκόρ 20% στο Κοινοβούλιο και 18,5% στη Γερουσία. Κάπως διαφορετικά έχουν τα πράγματα στις αυτοδιοικητικές εκλογές και τα αποτελέσματα εκεί. Εκεί η συμμετοχή είναι 26% στην εκπροσώπηση σε, στην τοπική αυτοδιοίκηση και ικανοποιούμεθα από το γεγονός ότι αυξάνεται ο αριθμός των γυναικών δημάρχων, κυρίως σε μικρές κοινότητες. Προέρχονται από την κέντρο αριστερά και την αριστερά ως επιτοπλίστων, αλλά ε, ως επιτοπλίστων δεν προέρχονται από κόμματα. Το 2010 οι εκλογές λοιπόν βελτίωσαν κατά τη την συμμετοχή των γυναικών. Δεν μπορούμε δηλαδή, θέλω να πω, να ακολουθήσουμε και να αρκεστούμε στις φυσικές εξελίξεις. Το 30% το όριο δεν το έχουμε υπερβεί ακόμα. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και θα πρέπει να το καταπιαστούμε διότι αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το γυναικείο μας δυναμικό. Μέχρι τώρα όμως το πρόβλημα δεν το εξέτασε κανείς, δεν κατέβαλε προσπάθειες και ο κυβερνητικός δεξιός συνασπισμός τα χειροτέρεψε τα πράγματα. Μια απόδειξη είναι το γεγονός ότι στο τωρινό ε, Υπουργικό Συμβούλιο δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα, ενώ λίγες είναι αναπληρώτριες υπουργοί, υφυπουργοί. Ε, έχουμε σχετικά πολλές γυναίκες στο κοινοβούλιο, σε ηγετικές θέσεις των δύο κοινοβουλίων, άνω κάτω βουλή, αλλά αυτό οφείλεται στις πιέσεις που ασκήθηκαν από την κοινωνία των πολιτών, γιατί πίεσαν για να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα. Θέλω να πω ότι αν θέλουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, χρειάζονται μέτρα για την πρόθεση της ισότητας των ευκαιριών. Χωρίς αυτά τα μέτρα θα βραδιπορούμε ή και δεν θα προοδεύουμε καθόλου. Δεύτερον, θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής πολιτική κουλτούρα παίζουν ρόλο στην εφαρμογή αυτών των μέτρων και παίζουν ρόλο θετικό. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν ιδιαίτερα την πρόεδρο τον, όχι, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Μπούζεκ και θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους άλλους που καταλαβαίνουν ότι όπως μια οικογένεια δεν πάει καλά όταν λείπει ένα βασικό μέλος, ο άνδρας ή η γυναίκα, έτσι δεν μπορούμε να έχουμε και λειτουργική ε, κοινωνία αν δεν συμμετέχουν οι γυναίκες στις ε, διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων. Χρειάζεται ένα θετικό κλίμα, μια κοινωνία όπου θα μπορούν να συμμετέχουν οι γυναίκες και θα δραστηριοποιούνται στην πολιτική. Για τη δημιουργία ενός τέτοιου κλίματος χρειάζονται εκδηλώσεις όπως αυτή. Στόχος μας είναι η ισότητα των ευκαιριών, η ίση μεταχείριση. Θέλουμε το, να αξιοποιήσουμε το δυναμικό ολόκληρης της κοινωνίας. Ευχαριστώ και πάλι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ευχαριστώ και την Επιτροπή Γυναικών και την Προεδρία του Συμβουλίου. Θα ήθελα να πω ότι είναι πάνω απ' όλα σημαντικές αυτές οι θετικές εμπειρίες οι οποίες θα πρέπει να παίξουν ρόλο για να βελτιωθεί και το κλίμα στη ζεχική Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η επόμενη ομιλητία είναι η Μαλένα Ρούπρεκτ, μέλον της Επιτροπής για Οικογενειακές Υποθέσεις τρίτη ηλικία τι γυναίκε και του νέους. Είναι από το Bundestag στη Γερμανία και θα τη δώσουμε μέσα στο λόγο. Παρακαλώ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμες συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ την Επιτροπή Γυναικών για την πρόσκληση με αφορμή την εκατοστή επέτειο της Διεθνούς ημέρας των Γυναικών. Για την ε, μέρα των γυναικών έγιναν στη Γερμανία πολλές συζητήσεις για την ε, ε, θέση ανδρών και γυναικών, ίσα δικαιώματα, ίση αμοιβή για ίση εργασία, για την εκπροσώπηση των, των, των γυναικών στην εργασία, στα χαμηλότερα αμοιβόμενα επαγγέλματα. Επίσης συζητήθηκε και η εκπροσώπηση των γυναικών στα Συμβούλια των Επιχειρήσεων. Τον Ιανουάριο του 2011 η πρώτη έκθεση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης με τίτλο «Ίσες ευκαιρίες στη Σταδιοδρομή ανδρών και γυναικών» δημοσιεύτηκε και εξετάζει τη συμμετοχή στην εκπαίδευση και στην ενεργό απασχόληση. Όλος τυχαίως η έκθεση αυτή δεν έτυχε της προσοχής της κοινή γνώμης, με την εξαίρεση κάποιες γυναίκες και τους πολιτικούς. Γι' αυτό σήμερα θέλουμε να συζητήσουμε για την ε, συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική. Ε, θέμα το οποίο παραμερίστηκε λίγο ε, στη Γερμανία εκτός και αν ένα ε, κόμμα συζητούσε συγκεκριμένα για ποσοστώσεις. Πώς ε, έχει το θέμα στην πραγματικότητα. Η καγκελάριος μας είναι γυναίκα. Πρώτη φορά στην ιστορία της Γερμανίας. Στη Γερμανία λέμε όμως ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Στην τωρινή κυβέρνηση με 14 υπουργού έχουμε 5 γυναίκες, δηλαδή η ποσόστοση έφτασε το 35%. Από 16 ομόσπονδα κρατήδια οι πρωθυπουργοί 2 είναι γυναίκες. Και αυτό πρόσφατη εξέλιξη είναι. Σε επίπεδο αυτοδιοίκησης η ποσόστοση είναι ακόμη χειρότερη. Τι γίνεται τώρα με τη συμμετοχή στα κόμματα. Από τα έξι κόμματα που εκπροσωπούνται στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, τρία έχουν στο καταστατικό τους ε, ποσοστώσεις, ρυθμίσεις για ποσοστώσεις. Και γι' αυτό έχουν και την υψηλότερη γυναικεία συμμετοχή, ποσοστό στο Κοινοβούλιο. Στο, εμείς οι σοσιαλδημοκράτες έχουμε 40-40-20 ποσόστοση, δηλαδή η ποσόστοση είναι 40% ε, για κάθε φύλλο και το 20% μπορεί να πληρωθεί από το ένα ή το άλλο φύλλο. Οι πράσινοι έχουν 50% ποσόστοση και η Λίνκε η Λίνκε, το κόμμα της αριστεράς πάλι το 50-50. Εδώ και λίγο καιρό έχει η Τσεντεού 25% και η Τσέσου το αδελφό κόμμα, το χριστιανοκοινωνικό κόμμα, συζητάει μήπως και εισαγάγει και αυτό ποσόστοση. Οι ελεύθεροι δημοκράτες, φιλελεύθεροι, δεν έχουν ποσόστοση στο Κοινοβούλιο και το αποτέλεσμα είναι ότι από τους 31 αυτό το κόμμα 23 είναι νέοι. Τώρα, τι νομικές προϋποθέσεις έχουμε στη Γερμανία. Από τον Ιανουάριο του 19 οι γυναίκες στη Γερμανία έχουν ε, δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε. Στο Σύνταγμά μας η συμμεταχείριση ε, ανδρών και γυναικών αναφέρεται στο άρθρο 3 όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το κράτος θα πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν και ό,τι απαιτείται για να εξασφαλιστεί η συμμεταχείριση. Τι γίνεται με την κοινωνία των πολιτών, τι γίνεται στην πολιτική. Εκεί πώς έχει το θέμα της ίσης μεταχείρισης. Οι ομάδες γυναικών και οι γυναίκες πολιτικοί που ασχολούνται με το θέμα βλέπουν ένα σοβαρό έλλειμμα. Γενικά αναγνωρίζεται το έλλειμμα, ε, κανείς δεν το αμφισβητεί πια, αλλά το αν απαιτούνται μέτρα για να λυθεί το πρόβλημα και να κλείσει αυτό το κενό που υπάρχει, εκεί διήστανται οι απόψεις και υπάρχουν έντονοι διαπληκτισμοί και αντιπαραθέσεις από οι νέοι άνδρες και οι γυναίκες τάσσονται στην πλειοψηφία τους κατά της ποσόστοσης θεωρώντας ότι οι επιδόσεις και τα προσόντα θα επιβληθούν. Αν ίσχυε αυτό θα έπρεπε τα τρία τέταρτα των κοινοβουλευτικών εδράνων να καλύπτονται από γυναίκες γιατί στη Γερμανία οι γυναίκες παίρνουν καλύτερους βαθμούς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην τριτοβάθμια και έχουν περισσότερα προσόντα. Άρα λοιπόν αυτό δεν ισχύει. Ζητώ λοιπόν το ε, ίδιο δικαίωμα ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών ε, και στα προσόντα. Ε, ζητώ να ε, διεκδικήσουμε το δικαίωμα να συμμετέχουμε ως γυναίκες ακόμα και με λιγότερα προσόντα ε, και όχι μόνο για αυτά. Τώρα, τι εμποδίζει την εφαρμογή της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης. Ε, νομίζω ότι η κατάσταση είναι παρόμοια σε όλη την Ευρώπη. Είναι αυτά τα παραδοσιακά μοντέλα, τα ταμπού, τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει ο άνδρας ή η γυναίκα στην κοινωνία, τι ρόλους πρέπει να αποδειχθεί. Άρα λοιπόν με βάση αυτά πολλές φορές δεν είναι εξασφαλισμένες και ανεξάρτητες οικονομικά παρά την καλή τους εκπαίδευση οι γυναίκες. Και οι ρόλοι προβλέπουν ότι πρέπει να κατανέμουν διαφορετικά και το χρόνο τους οι άνδρες και οι γυναίκες μεταξύ δουλειάς και φροντίδας όπως λέγεται. Από κανέναν άντρα ε, ο κανένας άνδρας δεν ερωτάται όταν ε, δραστηριοποιείται πολιτικά πώς λύνει το πρόβλημα των παιδιών, όπως ερωτήθηκα εγώ. Κανένας δεν τους ρωτάει ποιος θα φροντίσει τα παιδιά. Πολλοί είναι παντρεμένοι άνδρες ε, στο κοινοβούλιο και κανείς δεν τους ρωτάει τι θα τα κάνετε τα παιδιά σας. Τις γυναίκες όμως τις ρωτούν. Άρα λοιπόν έτσι διαμορφώνονται ρόλοι, πρότυπα και ε, διαμορφώνεται η κατανομή του χρόνου σε βάρος των γυναικών όταν είναι και γυναίκες και ε, έχουν οικογένεια και όταν είναι και μητέρες. Αυτή η διάκριση σημαίνει ότι οι ε, άγαμες και οι άτεκνες γυναίκες δραστηριοποιούνται στην πολιτική πιο εύκολα διότι δεν έχουν τα προβλήματα ε, της εγκυμοσύνης και όλα αυτά. Ένα άλλο πρόσκομα για μας είναι ότι η πολιτική είναι ανδροκρατούμενη σε ό,τι αφορά ε, την ε, διεξαγωγή της. Θεωρούμε ότι η οργανωτική δουλειά ε, οι άνδρες θεωρούν ότι η οργανωτική δουλειά γίνεται από κάποιους αφανείς ηρωές που φροντίζουν ε, τα πάντα στο σπίτι να εξασφαλίζεται η υποδομή άρα οι άνδρες μπορεί να ξενυχτήσουν σε συνεδριάσεις σε πολιτικές συγκεντρώσεις ενώ οι γυναίκες ε, δεν τα καταφέρνουν. Μια μεγάλη πρόκληση και μάλιστα έχουμε τη νέα Υπουργό μας για θέματα οικογένειας, η οποία τώρα ε, πρόκειται να γίνει μητέρα και είναι η μόνη υπουργό που ε, περιμένει παιδί. Και θα πρέπει βεβαίως να προβλέψει ε, χρόνο για να αναθρέψει το παιδί της που θα είναι τόσο μικρό. Ο άνδρας της που είναι πολιτικός δεν ερωτάται πώς θα συνδυάσει επαγγελματική ζωή και την ιδιότητα του νέου πατέρα. Παραδοσιακά πρότυπα λοιπόν, ταμπού και οι δομές που απορρέουν από αυτά σημαίνουν ότι φεύγουν από την πολιτική οι γυναίκες. Έγινε μια έρευνα για τις γυναίκες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μπορούσαν να συνδυάσουν και τα δύο ε, εργασία στην αυτοδιοίκηση και ε, ζωή στην οικογένεια. Ε, όταν γίνεται μια συνεδρίαση το βράδυ όπου η γυναίκα πρέπει να φροντίσει για το βραδινό φαγητό και να βάλει τα παιδιά για ύπνο, εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό πάλι οι γυναίκες κάνουν πίσω. Ο τρόπος εργασίας λοιπόν διέπεται από ανδρικά πρότυπα. Άρα οι γυναίκες απο, απορρίπτονται από αυτό τον τρόπο δουλειάς. Αυτό είναι καθαρό για μας πλέον. Ε, οι, οι γυναίκες αποθαρρύνονται από ε, τρόπο εργασίας αυτού του τύπου. Τι πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει να αλλάξουν και τα εκλογικά συστήματα για να ε, δούμε εάν δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος των γυναικών. Θα πρέπει να υπάρξουν ε, νομοθετικές ρυθμίσεις που θα προβλέπουν ε, ίσο χωρισμό του χρόνου ε, εργασίας και οικογενειακής ζωής για άνδρες και γυναίκες γιατί πολλές φορές επιβαρύνονται ιδιαίτερα οι γυναίκες επειδή θεωρείται ότι είναι πρικισμένες και ικανές και ε, αυξάνονται υπερβολικά οι απαιτήσει με αποτέλεσμα κάποια στιγμή ε, να ε, αποθαρρυνθούν. Οι διαφορές στην Ευρώπη είναι ελάχιστες. Η συμμεταχείριση από τον νόμο, από το Σύνταγμα έχει προχωρήσει αρκετά ε, στην Γερμανία δεν ε, ε, υπάρχει κανένας νόμος που να προβλέπει διακρίσεις. Άρα σε νομοθετικό επίπεδο έχουν επιτευχθεί πολλά. Στην πραγματικότητα όμως πώς θα επιτύχουμε την ίση μεταχείριση. Αυτό θα γίνει μέσα από μια εταιρική σχέση μεταξύ μας. Η ίση μεταχείριση και τα ίσα δικαιώματα βλέπω να γυρίζει πάλι ο θέμα στη, στις γυναίκες. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να δείξουμε μεγάλη υπομονή αλλά και να συνεργαστούμε με τους άνδρες ε, γιατί αλλιώς ε, θα χρειαστούμε περισσότερα χρόνια από το σαλιγκάρι στο κινέζικο τείχος για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στην πολιτική και στα κέντρα εξουσίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, και όλους τους εκπροσώπους από τα Εθνικά Κοινοβούλια και αμέσως τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Σύρπα Πιέτη Κέινεν, μέλος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επίσης μέλος της Επιτροπής των Δικαιωμάτων των Γυναικών και για την ισότητα και επιπλέον η κυρία Πιέτη Κέινεν έχει αναλάβει κάτι. Είναι η συγγήτρια για την έκθεση «Οι γυναίκες στην πολιτική». Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much for your kind words. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τις συναδέλφους για την πολύ σημαντική τους συμβολή για τις ιδέες τους. Για να είμαι σύντομη, πιστεύω πως η πολιτική, οι γυναίκες στην πολιτική είναι θέμα ποιότητας και ισότη, ισότητας και ποιότητας. Η ισότητα, καταρχήν πώς θα γίνει οι πληθυσμοί να έχουν τα ίδια δικαιώματα για να έχουν πρόσβαση ε, στους πόρους και στη λήψη των αποφάσεων. Και όταν ε, κάποιος μου λέει ε, ότι είναι κατά της πρόθεσης των γυναικών, των ποσοστών, των ποσοστώσεων μάλλον, Απαντάω πάντα ότι τότε θα έπρεπε να έχουμε και... Για σκεφτείτε μήπως έχουμε και ποσοστώσεις για τους πιο ηλικιωμένους λευκούς άνδρες. Ε, εγώ νομίζω πως η πολυμορφία δημιουργεί την ποιότητα στην λήψη των αποφάσεων. Έπειτα έχουμε αυτό το πολύ κρίσιμο τρίγωνο στην πολιτική, στις ανοιχτές κοινωνίες, δημοκρατία, συμμετοχική δημοκρατία, ευημερία ή σχετικά μικρές διαφορές εισοδημάτων και παιδεία. Αν κάποια από τις γωνίες του τριγώνου καταρρεύσει, ολόκληρο το κοινωνικό μας σύστημα θα καταρρεύσει. Και το είπε ήδη η κυρία Ρόμπινσον ότι οι κοινωνίε όπου υπάρχουν περισσότερε γυναίκε στη λήψη των αποφάσεων έχουν καλύτερη ισορροπία σε αυτό το τρίγωνο για την συμμετοχική διαδικασία, την καθολική παιδεία για όλου και την ευημερία για όλου. Ε, για μένα λοιπόν είναι θέμα ζωής και θανάτου να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στην λήψη των αποφάσεων. Μεγάλη διαφοροποίηση είδαμε τώρα από κράτος σε κράτος όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών ε, στο Κοινοβούλιο αλλά και στις κυβερνήσεις. Και αυτό είναι κάτι επί το οποίο θα πρέπει να δράσουμε. Και αυτή η έλλειψη ισορροπίας βλέπουμε να επικρατεί και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και αναφέρομαι στον αριθμό γυναικών, ε, στη... γυναικών επιτρόπων. Για το θέμα των διακρίσεων, έχουμε περισσότερες γυναίκες ε, στον κοινωνικό τομέα και στην εκπαίδευση σε σύγκριση με την κυβέρνηση και αν δει κανείς οριζόντια πόσες υπουργούς οικονομίας, οικονομικών έχουμε, θα εντυπωσιαστεί. Ακόμα και στις προοδευτικές χώρες, αν δει κανείς πόσες γυναίκες διατέλεσαν πρωθυπουργοί, υπουργοί οικονομικών, θα παρατηρήσει πως ε, τα νούμερα μειώνονται δραστικά. Τώρα, και στον ιδιωτικό και στον ε, δημόσιο τομέα θα πρέπει να προωθήσουμε τις γυναίκες όσον αφορά τη ε, διαχείριση των οικονομικών. Πολύ συχνά στην οικονομία Μιλάμε για επενδύσεις και για δαπάνες. Πολύ σημαντικές λέξεις αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ε, είναι και τώρα τελευταία και η λέξη πρόκληση. Για κάποιες φορές όταν χρησιμοποιούμε τα χρήματα για πιο συγκεκριμένες δράσεις Περισσότερο είναι στις, δαπα... στις επενδύσεις, ενώ όταν χρησιμοποιούνται τα χρήματα για, τον... Ε, για τους ανθρώπους συνήθως αφορούν δαπάνες. Κάτι άλλο που ήδη αναφέρθηκε εδώ είναι ότι έχουν λιγότερο, μικροχαμηλότερους πόρους συνήθως οι γυναίκες και η αντίληψη των μέσων μαζικής ενημέρωσης ε, τίνει να είναι διαφορετική όταν ε, ασχολείται με τις γυναίκες και τα θέματα των γυναικών από να αυτά των ανδρών. Και έπειτα υπάρχει και το θέμα της εμπιστοσύνης και θα έλεγα πώς θα δημιουργηθεί μια κρίτισιμη μάζα ώστε να εκτιμηθούν οι γυναίκες και η γνώμη των γυναικών. Χρειάζονται μεν ε, δράσεις, αλλά και νομοθεσία. Δράση, εγώ δεν έχω κάποιες απόλυτες απαντήσεις, αλλά υπάρχουν κάποιες καλές ιδέες που θα ήθελα να δούμε μαζί. Καταρχήν, πώς θα δημιουργηθεί η κρίσιμη μάζα και πώς θα υποστηριχθούν οι γυναίκες. Χρειαζόμαστε καλύτερα δίκτυα, διατομεακά και διακομματικά δίκτυα δίκτυα όπου διάφορες οργανώσεις γυναικών, η ΜΚΟ, θα συνεργάζονται όπου οι ηγέτες των συνδικάτων των πολιτικών κομμάτων, των επιχειρήσεων θα συναντώνται εκεί όπου τα, θα συζητώνται τα πολιτικά ζητήματα σε, πολιτικό, σε εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο η δυνατότητα δικτύωσης θα μπορούσε να βοηθήσει να ακουστούν οι φωνές και τα συμφέροντα των γυναικών. Χρειαζόμαστε Πιστεύω καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ πιο αποτελεσματική ε, στα εθνικά μας κοινοβούλια ή κατά τη διάρκεια των εκλογών, μην υποστηρίζοντας συγκεκριμένους υποψηφίους ε, ή πολιτικά κόμματα, αλλά δίνοντας τέτοια μηνύματα και βοηθώντας τις γυναίκες ε, να κάνουν την πολιτική τους εκστρατεία και να τονίσουν τη σημασία της εκλογής γυναικών. Και επίσης αναρωτιέμαι μήπως θα μπορούσαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουμε χωριστά προγράμματα για την κατάρτιση των γυναικών δημοσιογράφων ώστε να ασχολούνται περισσότερο με τα, με τα γυναικεία θέματα και την ισότητα των φύλων στην πολιτική. Τώρα, και την επόμενη φορά όταν θα ξανανοίξει η συνθήκη λόγω των οικονομικών ζητημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να θίξουμε και το θέμα των ποσοστώσεων ε, στους επιτρόπους. Γιατί πιστεύω ότι οι επίτροποι θα πρέπει να είναι μισή-μισή. Μισή άντρες, μισή γυναίκες. Κάθε κράτος μάλλον θα πρέπει να προτείνει έναν άνδρα και μια γυναίκα υποψηφίους, ώστε να διευκολυνθεί η κατάσταση και να φτάσουμε σε αυτή την ισορροπία. Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα και τις επιχειρήσεις, πιστεύω πως αν δεν δούμε εκεί σημαντική πρόοδο, το θέμα των ποσοστώσεων θα πρέπει επίσης να ληφθεί και εκεί υπόψη. Τελευταία μου τώρα παρατήρηση για τις νομικές δραστηριότητες και τα συνταγματικά δικαιώματα που θεσπίζουν ένα ισότιμο πεδίο για τις γυναίκες. Θα ήθελα λοιπόν να μπορέσουμε να δουλέψουμε καλύτερα, να δικτυωθούμε για να χρησιμοποιήσουμε αυτό το νέο στοιχείο ώστε να εξασφαλίσουμε και να εγγυηθούμε καλύτερη πρόσβαση των γυναικών στην πολιτική, όχι μόνο στα νούμερα, αλλά να εξαλειφθούν οι διακρίσεις γενικότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Πιέτη Κέινεν και ευχαριστήσω τους εθνικούς εκπροσώπους από Γερμανία, Τσεχία, Βέλγιο που κάνανε τις εισαγωγικέ παρουσιάσεις και έτσι μπορούμε να περάσουμε στην ε, συζήτηση. Όποιος επιθυμεί θα πάρει το λόγο. Η Ο Γιάννη Μπουντέν, συγγνώμη, είναι ο πρώτος στην ε, λίστα από την ε, Γαλλική Γερουσία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ που μου δίνεται για πρώτη φορά σήμερα το λόγο σε μια ανδρική φωνή. Χαίρομαι που έχουμε αυτή την ευκαιρία σήμερα που μας δίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να θίξουμε το, το ρόλο των γυναικών στην ευρωπαϊκή πολιτική. Διότι, διότι τα μαθήματα που μπορούμε να τλήσουμε από τις εθνικές μας εμπειρίες αποτελούν ένα μοχλό θα λέγαμε για να προχωρήσουμε σε ένα τομέα ο οποίος είναι σημαντικός για την, το μέλλον της δημοκρατίας οι γυναίκες ε, αποτελούν το μισό και κάτι παραπάνω του πληθυσμού. Και σήμερα βλέπουμε, ε, διαψώνουμε απλώς ότι αποτελεί ένα πρόβλημα η μικρή τους παρουσία στα διάφορα θεσμικά οργανά. Εγώ εκπροσωπώ τη Γερουσία, είμαι από τη Γαλλία και πραγματικά δεν μπορώ να πω ότι χαίρομαι με την κατάσταση παρόλο που είχαμε μια πρόοδο και 10 χρόνια, όπως το είπε εξάλλου και η κυρία Προλαλήσασα. Ε, πραγματικά δεν βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλή θέση όσον αφορά τη θέση των γυναικών στην πολιτική σε σχέση με την παγκόσμια κλίμακα. Ε, και βρισκόμαστε μάλιστα στην 73η θέση όταν βλέπουμε τα εθνικά κοινοβούλια. Με 23,5% στην παρουσία γυναικών στην ε, στη Γερουσία, ενώ μόνο 18% έχουμε στην Εθνοσυνέλευση. Αυτό σαν παρηγοριά για μας. Η Γαλλία, ε, παρόλα, παρόλα αυτά να θίξω ότι ε, άργησε να δώσει το δικαίωμα για ψήφους στις γυναίκες το 1940. Το 2000 με τον Πρωθυπουργό των τον Ζωσπέν, γίνανε κάποιες αλλαγές. Ε, είχε γίνει μια αλλαγή ήδη το 1999 στο Σύνταγμα, όπου ο νόμος δίνει μια ίση εκπροσώπηση ανθρώπων γυναικών στην, ε, στα διάφορα εκλέξιμα όργανα. Υπήρξε συζήτηση στο Κοινοβούλιο για το νόμο αυτό του 2000 που επιβάλλει μια ισότητα ανδρών γυναικών. Ο μηχανισμός που πέρασε με αυτό τον νόμο επέτρεψε στην ισότητα κατά κάποιο τρόπο να γίνει πράγματι μια πραγματικότητα. Αυτό το είδαμε σε ορισμένες ε, συνελεύσεις αλλά όχι σε όλες. Υπήρξε πρόοδος ε, όπου έχουμε ε, λίστα στις εκλογές όπου προβλέπεται ότι όλες οι λύσεις θα πρέπει εναλλακτικά να αποτελούνται από έναν υποψήφιο από κάθε φύλλο. Το βλέπουμε αυτό στα περιφερειακά συμβούλια, όπου έχουμε 48% παρουσία γυναικών και με 40% ήδη εκπρόσωποι, ε, εκπροσωπούνται στα συμβούλια αυτά ε, οι αντιπροεδρίες από γυναίκες. Επίσης βλέπουμε ότι αυτό ισχύει στα δημοτικά συμβούλια όπου βλέπουμε και εδώ μια παρουσία 40% το εκπροσώπηση μάλλον των γυναικών. Επίσης στην ευρωπαϊκή εκπροσώπηση εδώ στο Ευρωπαϊκό Γενοβούλιο βλέπουμε από το 2009 και μετά έχει πάνω από 40% εκπροσώπηση στο γενικό φύλλο. Αλλά αυτές οι μηχανισμοί ε, ε, ισχύουν μόνο σε εκλογές που γίνονται με λίστα. Όπου έχουμε ε, εκλογές με δύο γύρους, ε, τα αποτελέσματα είναι απογευτευτικά πολύ χαμηλό το ποσοστό γυναικών στα... Ε, ε, έχουμε την εκπρόσωψη γυναικών στα νομαχιακά συμβούλια. 18% γυναικών στην Εθνική Σύνεθνο Συνέλευση. Οι διατάξει που υποτίθεται γίνανε από τα κόμματα για να προωθήσουν τη θέση των γυναικών πραγματικά δεν πετύχαν τίποτα. Ακόμα και όταν υπάρχουν κυρώσει οικονομικές στα κόμματα, διότι δεν παρουσιάζουν αρκετέ ε, υποψήφιε στι εκλογές ή ακόμα και όταν έχουμε ένα κανόνα για το πώς εκπροσωπείται κανείς στα καντόνια ε, και ε, το αν θα αντικατασταθεί όχι από άτομο του άλλου φίλου Πέρα από όλου αυτούς του ε, περιορισμούς δεν έχουμε κανένα σωστά αποτελέσματα. Γι' αυτό παρορούμε να πούμε ότι σήμερα το θέμα της ισότητας η γυναίκα είναι κάτι το οποίο μένει να γίνει. Βλέπω την πρόοδο ότι έχει επιτευχθεί, όπω είπα, μόνο σε εκλογέ οι οποίε γίνονται με λίστα. Για, κατά τα άλλα, ε, η θέση των γυναικών είναι επισφαλή. Και η συνάδελφό μου, Κατρίν Μορέν, αφήνω σε αυτή να, να αναφερθεί στην υποχώρηση που γίνεται όσον αφορά την πρόσβαση γυναικών ε, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. παρόλη την νομοθεσία που ε- εγκρίθηκε την περασμένη χρονιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στην επόμενη εκπρόσωπο, εκπρόσωπο από την Γερουσία και αυτή της Γαλλίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, βλέπετε η Γαλλική Γερουσία παρουσιάζεται ενώπιον σα με τον πιο ισότιμο ε, τρόπο που μπορούσε, γιατί ταυτόχρονα βλέπετε έναν αντιπρόεδρο και μια αντιπρόεδρο της, ε, της Επιτροπής για τα Δικαιώματα της Γυναίκας που συμμετέχουμε σε σημερινή συνεδρίαση. Ο συνάδελφος μου δεν σας ε, παρουσίασε μια εικόνα της ισότητας στη γυναίκα και των μηχανισμών που την ευνόησαν. Και φυσικά αυτό βασικά οφείλεται στον κανόνα που επιβάλλει στις εκλογές που γίνονται με βάση λίστες, εκλογικές λίστες που επιβάλλει έναν υποψήφιο από κάθε φύλλο. Οι πρόοδοι που οφείλονται σε αυτόν τον μηχανισμό είναι σημαντικές αλλά τελείς. και βέβαια η ισότητα έχει προχωρήσει στις εκλογές που γίνονται με βάση εκλογικές λίστες. Δυστυχώς στις εκλογές που γίνονται με την πλειοψηφία και με επιλογή μόνο ενός ονόματος ε, οι πρόοδοι είναι πολύ ευάλωτες και μια αλλαγή μπορεί να αμφισβητήσει. Η νέα εκλογή μάλλον μπορεί να αμφισβητήσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί εκεί. Παρ' όλα αυτά οι νομοθεσίες που ε, υιοθετήθηκαν πέρσι δίνουν ένα σαφές παράδειγμα. Εδώ δεν θα σας μιλήσω για τις μεταρρυθμίσεις για, τις ε, για, για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλουμε για τους περιφερειάρχες και τους νομάρχες να αντικαταστήσουν από, ε, από εκπροσώπους που θα εδρεύουν και στα νομαρχιακά και στα περιφερειακά συμβούλια. Η απειλή τώρα είναι ότι θα γίνει αυτό και για τις εκλογές που θα γίνουν για αυτούς τους, τους ε, δαφικούς ε, συμβούλους. Η κυβέρνηση επέτρεψε ε, θα πρέπει να ομολογήσουμε τη δημιουργία μιας γνήσιας ε, ισότητας και θεώρησε ότι θα πρέπει να γίνει η... γίνουν οι εκλογές με δύο γύρους, πράγμα το οποίο βέβαια ε, ευνοεί την, την εγκύτητα αλλά δεν επιτρέπει να γίνει σεβαστή η, σεβαστός ο πλουραλισμός ούτε η ισότητα. Για να σας το θυμίσω με αυτό το είδος των εκλογών μόνο 12% είναι οι νομάρχες γυναίκες Επίσης, στη Γερουσία ασχοληθήκαμε με το θέμα και φτιάξαμε μια ανέκθεση με την, η οποία φέρει τον τίτλο «Πρέπει να σωθεί η ισότητα» και που διατυπώθηκαν διάφορες συστάσεις που υιοθετήθηκαν ομόφανα από τα μέλη της Γερουσίας, από όλα δηλαδή τα πολιτικά κόμματα. Διερωτηθήκαμε σε ποιο βαθμό ένα τρόπο εκλογή που θα υποβαθμίσει την ισότητα μπορεί να συμφιλειωθεί με τον συνταγματικό στόχο, τον νόμο δηλαδή, που ευνοεί την ίση πρόσβαση γυναικών και ανδρών στον εκλογικό κόσμο και στη ερετά αξιώματα. Ε, δεν θέλουμε βεβαίως να περιορίσουμε την ελευθερία του Κοινοβουλίου όσον αφορά τον εκλογικό νόμο, αλλά αυτή η ελευθερία θα πρέπει να πλήξει με άλλους τρόπους τον συνταγματικό ε, στόχο της ίσης πρόσβασης. Επίσης δεν ευνοήσαμε τον οδό των οικονομικών κυρώσεων που επιβαλήθηκαν στα κόμματα για να τηρήσουν την ισότητα, γιατί θεωρήσαμε ότι τελικά δεν είχαν και αντίκτυπο. Η προώθηση, το, μάλλον η αντιστοιχεία, η αναλογία των γυναικών στην ε, γαλλική πολιτική ζωή μας κάνει να αμφισβητούμε το κέρδος. Ωστόσο, κοστίζουν ε, στα κόμματα 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο τα μέτρα αυτά. Τώρα, σε κάθε περιοχή οι εκλογές προτείνουμε να γίνει από, με βάση μια διπλή επιλογή, δηλαδή έναν άνδρα και μια γυναίκα υποψηφίους. Ε, έτσι θα μειώσουμε κατά το ίμιση τον αριθμό των περιφερειών που έχουν οριστεί για την εκλογή τους. Η εφαρμογή ενός τέτοιου τύπου εκλογικού νόμου θα επέτρεπε να καθοριστεί αυστηρά η ισότητα. Θα είχε επιβληθεί. Βεβαίως είναι πολύ καινοτόμα αυτή η ιδέα, δεν εγκρίθηκε, αλλά πιστεύω πως στο μέλλον θα πρέπει να εμβαθύνουμε σε αυτή την ιδέα και γι' αυτό και ήθελα να την μοιραστώ μαζί σας. Τέλος, να σας αναφέρω κάτι ακόμα σημαντικό, γιατί η προσωπία μας ασχολήθηκε φέτος με τη τους ε, όρους, τις συνθήκες που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την ισότητα στην πολιτική ζωή αλλά και στην επαγγελματική ζωή και κροαστήκαμε στο πλαίσιο των εργασιών μας και αναθέσαμε στη κυρία Ράιζερ να εκπονήσει μια έκθεση. Ο Υφυπουργό Ισότητα ε, Βαλερή Λετά ζήτησε την εκπόνηση αυτή τη έκθεση και αυτή αποδεικνύει ότι τελικά στι τηλεοπτικέ μα οθόνε, αντίθετα με το τι μπορεί να σκεφτόμαστε, η εικόνα ε, τη γυναίκα συχνά είναι στερεότυπη και ανεπαρκή. Εν γέννη, οι γυναίκε αντιπροσωπεύονται πολύ λιγότερο από ότι οι άνδρε και αν ε, αντιπροσωπεύονται, είναι συνήθω σε ρόλους δευτερεύοντες ε, θύματος ή μάρτυρα, ποτέ σε ρόλους ε, πυρογνωμόνων επαγγελματιών. Και σας προτείνω σε όλους να δουλέψουμε στους στόχους για τη δημόσια τηλεόραση, ε, να δουλέψουμε υπέρ μιας πιο ευνοϊκής γυναίκας για τη, εικόνα συγγνώμη, για τη γυναίκα, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την ισότητα. Πρόεδρος. Eh, Ευχαριστώ. Τώρα θα δούμε τι ακριβώς ισχύει στη Λιθουανία. Η κυρία Χάιλον ναι, θα μας ενημερώσει για αυτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι μαζί σας ε, σήμερα το πρωί για να συζητήσω την έννοια της Διεθνούς ημέρας της γυναίκας που άλλαξε τον κόσμο. Αναλογιζόμενοι το μέλλον του πολιτικού ρόλου της των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούμε ότι ο ρόλος αυτός πρέπει να αναβαθμιστεί σε σημασία. Θέλουμε περισσότερες γυναίκες στη, στα κέντρα λήψης αποφάσεων, περισσότερες γυναίκες αρχηγούς όμως ε, οι γυναίκες ε, ε, διαφορετικά εκπροσωπούνται στα πολιτικά κόμματα. είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν οι ποσοστώσεις για να εντοπίσουν και να προωθήσουν προσωπικότητες γυναικών. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ε, εστίαση σε γυναίκες προκισμένες με μια ε, διεθνή ή μεγαλύτερη εμβέλεια. Δεν είναι δεν μπορούν να κατανοήσουν βαθιά όλες οι γυναίκες πολιτικοί τα θέματα του φύλου, της ταυτότητας των φύλων, τα ανθρώπινα δικαιώματα τα γυναικεία θέματα όπως δικαίωμα αναπαραγωγής, οικογενειακός προγραμματισμός, ε, εκπαίδευση σεξουαλικότητας, ε, εκπαίδευση σεξουαλικών μειονοτήτων κλπ. Πιστεύω λοιπόν ότι στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τονίσουμε περισσότερο την ε, ανάδειξη της προσωπικότητας της γυναίκας, της αυτοπεποίθησης, της εκπαίδευσης της γυναίκας, της ψυχολογικής ευελιξίας της γυναίκας, της ευθύνης, της αφοσίωσης της γυναίκας. Ο πολιτικός φεμινισμός αρχίζει στα πολιτικά κόμματα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου γυναίκες στα πολιτικά κόμματα χάνουν το ατομικό τους πρόσωπο και γίνονται φερέφωνα της κομματικής ιδεολογίας. Όταν οι γυναίκες περνούν την συντηρητική ιδεολογία, τη στερεοτυπική, τη δογματική αντίληψη των συντηρητικών κομμάτων, καταστρέφουν τις ίσες ευκαιρίες και την πολιτική της ισότητας των φύλων. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι αλληλέγγυες, όχι κατακαιρματισμένες. Πρέπει γι' αυτό να αλλάξει η γυναικεία νοοτροπία. Θα πρέπει οι γυναίκες να διαμορφωθούν σε προοδευτικές προσωπικότητες που θα συνδυάζουν, θα συνδέουν το σύστημα των ποσοστώσεων αφενός με μια ιδιαίτερη σημασία στην ανάδειξη και διαμόρφωση της γυναικείας προσωπικότητας. Ευχαριστώ. Τώρα θα δούμε πώς έχει η κατάσταση στην Πορτογαλία. Η κυρία Μαρία Ντορσάιρο Κανάιρο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, ήδη αναφέρθηκε επανελειμμένος ότι η ισότητα των φύλων είναι παράβατο ανθρώπινο δικαίωμα, είναι, θέμα, είναι αξία δημοκρατική και θα πρέπει να υποστηρίζεται. Στην Πορτογαλία εμείς το 2006 θεσπίσαμε το νόμο περί που εισάγει την ποσόστοση 33% παρουσία της ομάδας που υποαντιπροσωπεύεται στις εκλογικέ λίστες ώστε να, υπάρξουμε, να, να πετύχουμε μια πιο ισορροπή εκπροσώπηση των γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων. Είναι προφανές ότι αυτό το μέτρο σε συνδυασμό με άλλα μέτρα που λήφθησαν όπως εκείνο που προκύπτει από το Ναστικό κώδικα για την, τον συνδυασμό της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή και διάφορες δομές αλλά και το εθνικό πρόγραμμα για την ισότητα που προβλέπει μηχανισμούς ε, ε, για την διευκόλυνση της συμμετοχής των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων πετύχαμε λοιπόν αποτελέσματα που τελικά οδήγησαν στην συμμετοχή των γυναικών, περισσότερων γυναικών μάλλον, στο Ευρωκοινοβούλιο. Είμαστε κοντά στο 35% και, και στους Δήμους όπως ήδη αναφέρθηκε στο πρώτο τμήμα της συζήτησης, ήμασταν αρκετά χαμηλά, είμαστε στο 20% περίπου και ορισμένες φορές, σε ορισμένες περιπτώσεις, σπανίως φτάνουμε μόνο στο 10%. Αυτός ο βασικός μηχανισμός για την εγγύηση της πιο ισότιμης εκπροσώπησης των γυναικών στα μέσα ε, της εξουσίας στην ουσία προκύπτει από μια απλή χρήση ποσοστώσεων. Η Γαλλία είπε ότι η νομοθεσία σχετική επιβάλλει έναν κανόνα εναλλαγή, δηλαδή έναν από το κάθε φύλλο. Εμείς λέμε τρεις και τρεις, γιατί μόνο σε δύο λίστες ε, βλέπουμε να υπάρχουν ε, πρώτα οι γυναίκες, ε, πράγμα που σημαίνει ότι τελικά Εμείς επιτύχαμε τον τελικό στόχο που ήταν 33%. Ε, και στην κυβέρνηση δεν υπάρχει, δεν έχει εφαρμοστεί ο κανόνας των ποσοστώσεων. Τώρα βέβαια φαίνεται πως τελικά υπήρξε θετικός αντίκτυπος γιατί φτάνουμε και εκεί στην εκπροσώπηση κατά 20%. Όπως ήδη αναφέρθηκε στο πρώτο κομμάτι της συζήτησης, το θέμα της ισότητας ή της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα όργανα Τη πολιτική εκπροσώπηση θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα και σε άλλα όργανα λήψης αποφάσεων όπως στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων, σε ερευνητικά συμβούλια και ούτω καθεξής. Και εγώ αναφέρομαι στην κατάσταση της χώρας μου. Δεν υπάρχει καμία γυναίκα σε κανένα οικονομικό θέμα, χαρτοφυλάκιο. Καμία γυναίκα στη διοίκηση της κεντρικής μας τράπεζας και στις 20 καλύτερες επιχειρήσεις Μόλις 4% είναι οι γυναίκες και όταν είδαμε ποια είναι η παρουσία των γυναικών ας πούμε στους ε, διευθυντές πανεπιστημίων, στους πριτάνες και τα λοιπά δεν φτάσαμε ούτε στο 5%. Γι' αυτό και τίθεται αυτό το θέμα της αύξησης της συμμετοχής. Είναι επιταγή αυτό της βιώσιμης ανάπτυξης. Και θα πρέπει οι ποσοστώσεις να συνδυαστούν με άλλα μέτρα δεν μπορούμε να επιβάλλουμε ποσοστώσεις στον ιδιωτικό τομέα, αλλά τουλάχιστον ε, θα πρέπει να σκεφτούμε κάποια κίνητρα ώστε ο ιδιωτικός τομέας να θεωρήσει ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα εξέλιξης μέσω κυρώσεων, μέσω ε, ποιών μέτρων, πιο βολονταριστικών μέτρων στη συμμετοχή γιατί το κόστος αυτής της ε, έλλειψης ισορροπίας στα όργανα αποφάσεων ε, στα διάφορα επίπεδα είναι πολύ ψηλό γιατί ε, και αβάσταχτο πολλές φορές για την ανάπτυξη των κοινωνιών από την άποψη της δημοκρατίας αλλά και από την άποψη της ανάπτυξης. Και εγώ να σας αναφέρω μόνο δύο παραδείγματα που τουλάχιστον στη χώρα μου έχουν τεράστιο κόστος από την άποψη της ε, εξέλιξης, δηλαδή συνέπειες δημογραφικές και οι αλλαγές της συμπεριφοράς. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να είμαστε πιο δημιουργικοί, πιο αποφασιστικοί και να σκεφτούμε μια πολιτική σε μια τέτοια συγκυρία όπου σίγουρα δεν είναι θετική για την βιωσιμότητα της ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Η επόμενη παρουσίαση είναι από τη Σλοβακία. Άννα Μπελόρτσοβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να δώσω κάποια στοιχεία για το θέμα αυτό. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα, τη Σλοβακία, όπου στο άμεσο μέλλον δεν προβλέπεται εισαγωγή ποσοστώσεων. Μια χώρα όπου το πολιτικό κόμμα στην εξουσία απορρίπτει τις ποσοστώσεις, απορρίπτει και συγκεκριμένο ποσοστό γυναικών στο ψηφοδέλτιο. Τώρα είναι 16% το ποσοστό στο Κοινοβούλιο των Γυναικών. Άκουσα την κυρία από την Ελλάδα που είπε ότι πέτυχαν 17% με ποσοστώσεις. Άρα εμείς έχουμε επιτυχία. Παρόλο που για πρώτη φορά έχουμε πρωθυπουργό γυναίκα, στα πρώτη φορά στην ιστορία της Σλοβακίας, δεν βελτιώθηκε όμως από εκεί η συμμετοχή των γυναικών, γιατί εκτός από την πρωθυπουργό Μία μόνο γυναίκα υπουργό βρίσκεται μεταξύ όλων των ανδρών που Είναι όμως υπουργό δικαιοσύνη. Τώρα, εκπροσώπηση στο Σλοβακικό Κοινοβούλιο. Η εκπροσώπηση είναι μικρή, αλλά από την άλλη πλευρά, ε, επειδή έχουμε το σύστημα της αναλογικής και καμιά φορά η σταθερότητα της κυβέρνησης μπορεί να ε, εξαρτάται και από δύο ε, ψήφους στο Κοινοβούλιο. Είναι πολύ προσεκτικοί όταν τοποθετούν στο ψηφοδέλτιο μια νέα γυναίκα γιατί σκέφτονται το ενδεχόμενο της ε, εγκυμοσύνης που θα την διώξει από το Κοινοβούλιο. Το Σύνταγμά μας λοιπόν περιορίζεται να πει ότι η ε, εντολή δεν προβλέπει άδεια μητρότητας ε, ή γονεϊκή άδεια για μέλος του Κοινοβουλίου. Οπότε θα πρέπει η γυναίκα αυτή, αν καταστεί έγκυος, να παραιτηθεί. Κάτι ακόμα που αφορά το πρώτο μέρος της ε, σημερινής εκδήλωσης. Στη Σλοβακία υπάρχει ο λεγόμενος, ε, ε, η, λεγόμενος, η λεγόμενη πρωτογενής ψήφος, ε, δηλαδή θα πρέπει να συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος 3% όλων των ψήφων που πηγαίνουν σε αυτό το πολιτικό κόμμα για να εισέλθει στο Κοινοβούλιο. Ερωτώ λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να δοθούν περισσότερες τέτοιες προτιμησιακές ψήφοι στις γυναίκες γιατί αν η γυναίκα είναι ας πούμε πεντηκοστή στη, στο ψηφοδέλτιο, αλλά αν, ψηφισ... αν όλες οι γυναίκες που θα έρθουν να ψηφίσουν τις εξασφαλίσουν ψήφο, τότε θα ανέλθει στην πρώτη εκλόγιμη θέση. Γιατί οι γυναίκες, δηλαδή ερωτώ, δεν εκλέγουν γυναίκες πέρα από τα προσόντα του υποψηφίου. Πολύ συχνά δεν ψηφίζουν οι γυναίκες γυναίκες. Πολύ συχνά οι γυναίκες δεν θεωρούν τις γυναίκες αρκετά ικανές και ε, ότι δεν έχουν αρκετά προσόντα και ψηφίζουν άντρες. Γιατί δεν μπορεί να αλλάξει λοιπόν αυτό. Επίσης, ε, μιλήσαμε πολύ για ποσοστώσεις. Θέλω να σας ρωτήσω πού είναι η εγγύηση ότι οι ποσοστώσεις θα επιφέρουν και ποιότητα στην πολιτική. Πού στο αποσκοπεί η ποσόστοση, απλώς ε, να επιτύχει ένα ποσοτικό στόχο ότι μάλιστα εκλέξαμε τόσες και τόσες γυναίκες. Εμείς σήμερα γιορτάζουμε τα 100 χρόνια των αγώνων των γυναικών για τις ελευθερίες και τα δικαιώματά τους. Από την άλλη πλευρά, καμιά φορά μου φαίνεται ότι οι αναπτυγμένες χώρες ε, οφείλουν πάρα πολλά ακόμη στις γυναίκες. Δεν έκλεισε το κενό στις αμοιβέ. Δεν λύθηκε το πρόβλημα της βίας. Δεν μιλάμε μόνο για τη θέση των γυναικών στον Ισλαμικό κόσμο. Δείτε και εδώ τι γίνεται. Σε πολλές δημοκρατικές χώρες ε, υπάρχουν προβλήματα. Πόσες και πόσες ακόμη δεν πέφτουν θύματα ε, βία στο σπίτι. Ας κοιτάξουμε λοιπόν τα του οίκου μας επίσης και Επίσης μιλάμε ξανά και ξανά για τη φροντίδα των παιδιών. Αυτό πάντα θα, συνεχί... θα, είναι ε, ε, θέμα γυναικών. Σήμερα βλέπουμε ότι πολλές γυναίκες αναβάλουν να γεννήσουν παιδί ε, παρά μόνο αφού περάσουν τα 30. Πολλές φορές δηλαδή πιέζονται να αντιμετωπίσουν το δίλημα στα βιοδρομία ή οικογένεια. Και αυτό δεν είναι δικό τους δίλημα, ε, ε, δηλαδή δεν το προκαλούν εκείνες, αλλά η κοινωνία που δεν προσφέρει στις νεαρές αυτές γυναίκες αρκετές δυνατότητες και τις πιέζει να, ε, να αναγκαστούν να διαλέξουν στα διοδρομία οικογένεια. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί δεν εκπροσωπούνται στην πολιτική οι γυναίκες. Δεν είναι απλή απάντηση δεν ε, ε ναι, λύνεται το πρόβλημα με τις που είναι και λίγο προσβλητικές ε, θεωρώ γιατί θα πρέπει για να δούμε γιατί δεν ε, συμμετέχουν στην πολιτική αρκετές γυναίκες να δούμε τις ρίζες του προβλήματος, τα πραγματικά αίτια και να μπούμε σε μια διαδικασία ένταξής τους και προσέλκυσής τους. Ας ε, στηρίξουμε λοιπόν τις γυναίκες στη ζωή τους στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν μπορούν να εκπροσωπούνται αρκετά. Περίμενα στη σημερινή εκδήλωση να επικεντρωθούμε όχι μόνο στις γυναίκες στην πολιτική αλλά γενικά στις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, στις γυναίκες τις οποίες η κοινωνία εξακολουθεί να οφείλει ακόμη πολλά. Και ένα τελευταίο σχόλιο που αφορά κάτι που είπε ο κύριος Μπούζεκ ότι ακόμα και όταν μιλάμε για την ισότητα μην ξεχνάμε ότι είμαστε γυναίκες και ο κύριος Μπούζεκ μας συνεχάρει με αφορμή την επέτειο της Διεθνούς ημέρας της γυναίκας αλλά Νομίζω ότι θα ξύζαμε και ένα λουλούδι από εκείνον. Δηλαδή τις γυναίκες της... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η επόμενη ομιλητή ομιλήτρια είναι η Βόνα από την Πολωνία. Ε, γεια σας κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ που έχω τη δυνατότητα να είμαι εδώ μαζί σας είναι ένα θέμα ε, στο οποίο μπορούμε όλοι από κοινού να αγωνιστούμε για να λύσουμε πολιτικά προβλήματα. Δεν υπάρχει καμιά χώρα όπου οι γυναίκες είναι ευχαριστημένες. Ο πρόεδρος έκανε μια εισαγωγή και είπε πράγματα ενδιαφέροντα. Τώρα, η πρωτοβουλία από αυτήν την ομάδα με συνάντηση με τα μέλη και έγινε μια συνάντηση τον Ιούνιο ε, στη Βαρσοβία και μετά είχαμε και το Δεκέμβριο του 2010 ε, που αποφασίστηκε ε, σε μας ένα πρόγραμμα, μια πρόταση για ε, δικαιώματα, ε, να αλλάξει ο νόμος για να υπάρχουν ίσα δικαιώματα για των γυναικών σε όλες τις ε, εκλογές. Εγώ το θεώρησα αυτό πάρα πολύ θετικό, όπως καταλαβαίνετε. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να, ακούσουμε, να ακούμε μάλλον και το τι ακριβώς γίνεται στις άλλες χώρες. Τον Ιανουάριο στην Πολωνία είχαμε νομοθεσία η οποία ίσως να μην είναι καταπληκτική, αλλά ε, όσον αφορά το θέμα της ισότητας κατά 50% αλλά παρά αυτά αποτελεί ένα πρώτο βήμα θα έλεγα αυτό με τις ποσοστώσεις. Φτάσαμε στο επίπεδο 35% της ποσοστήσης. Αλλά δεν, δηλαδή δεν θα, υπάρχει, δεν θα επιτρέπεται να υπάρχει μικρότερο ποσοστό εκπροσώπησης γενικών σε ένα κατάλογο υποψηφιωτήτων. και όταν έχουμε να κάνουμε μια λίστα η οποία δεν εκπληρώνει αυτούς τους όρους, περνάει, τη στέλνουμε σε μια επιτροπή η οποία πρέπει να ε, ελέγξει, ζητούν μια διορθωτική κίνηση και αν αυτό δεν γίνεται, τότε η Επιτροπή για τις εκλογές μπορεί να απορρίψει κάτι, μια τέτοια λίστα. Στην ακραία περίπτωση τώρα αυτό λέμε. δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αφού ε, περάσαν αυτές οι ποσοστότητες γιατί θα είμαστε για πρώτη φορά σε μια τέτοια κατάσταση και θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργούν τα πράγματα. Το ε, φθινόπωρο μάλιστα που θα έχουμε εκλογές για το κοινοβούλιο τότε θα το δούμε. Αυτό είναι λοιπόν ένα βήμα στο δικό μας αγώνα ε, για τον αγώνα για την ισότητα. Φυσικά όμως ε, δεν λύνονται όλα τα προβλήματα έτσι. Το καλύτερο θα ήταν είναι να ξεπεράσουμε αυτό το θέμα ε, και να μπορέσουμε να σιγουρέψουμε θέσεις. διότι έτσι δεν εξασφαλίζεται η παρουσία γυναικών στο κοινοβούλιο. Όπως καταλαβαίνω. Δηλαδή μπορεί να εξασφαλίσει κανείς με την ποσόστοση της υποψηφιότητες, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα περάσουν και στη ε, εκλογή. Δεν είναι δηλαδή μια σίγουρη ε, επιλογή ε, για να υπάρχει μεγαλύτερη εκπροσώπηση γυναικών ή τι η ποσόστοση δεν είναι η καλύτερη λύση. Θα πρέπει δηλαδή να διασφαλιστούν και θέσεις εκλέξιμες. Ε, λοιπόν, να μην πω στατιστικά τώρα για να σας πω πώς ακριβώς έχει η θέση των γυναικών. Δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Ε, έχει βελτιωθεί το επίπεδο εκπαίδευση, αλλά στα σημαντικά πόσα δεν έχουμε ε, πολλές γυναίκες σε υψηλά, σε υψηλές και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπρόσωψη δεν είναι καλή θα έλεγα ικανοποιητική. Κυρίως άνδρες ε, εκπρόσωπουν την Πολωνία. Ίσως όμως αυτή η νομοθεσία που σα ανέφερα να οδηγήσει σε κάτι τέτοιο να έχουμε καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών. Τώρα, για τη θέση των γυναικών στην Πολωνία. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε κάποια ικανοποιητική κατάσταση οι νέες γυναίκες ε, όταν θέλουν να ζητήσουν μια δουλειά αμέσως ρωτάνε αν θέλουν, αν σκοπεύουν άμεσα να ε, δημιουργήσουν οικογένεια. Ε, τέτοια ερωτήματα δέχονται. Και συχνά δεν αποκτά κανείς την θέση εργασίας Κάτι που το οποίο δεν ισχύει για τον άνδρα, γιατί όπω καταλαβαίνετε ο εργοδότη σκέφτεται πάντοτε το θέμα της ε, αδεία που θα, που θα ακολουθήσει μετά από μια γένα και τα παρεμφερεί. Έχουμε πέντε γυναίκες υπουργού στην κυβέρνηση τη Πολωνία. Σω να μην είναι και τόσο άσχημο σε σχέση με άλλε χώρε. Πέντε γυναίκε υπουργοί, κάτι είναι και αυτό. Αυτό θετικό θα μπορούσα να πω ότι είναι. Τώρα, γιατί δεν ε, ε, στρατεύονται στο πολιτικό στίβο θα λέγαμε οι γυναίκες. Διότι υπάρχει το θέμα του κινήτρου. Ε, από τη μικρή ηλικία μεγαλώνοντας δεν διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο να υπάρχουν και ανάλογες φιλοδοξίες και επιδιώξεις. Υπάρχουν φυσικά και τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη φροντίδα των παιδιών αλλά το σημαντικότερο θα έλεγα πρόβλημα είναι να αλλάξει η στάση, η οπτική γωνία των ανδρών. Ο τρόπος που σκέφτονται. δεν δέχονται και δεν έχουν και κίνητο, δεν παροτρύνονται από, τους, ε, από το θα λέγαμε. Αν δεν αλλάξει και όσο δεν αλλάζει θα έλεγα η οπτική γωνία από την πλευρά των ανδρών, όσο θα είναι δύσκολο να αλλάξει η θέση των γυναικών. Και τέλος να ευχηθώ ε, όλες τις γυναίκες ε, καλή επιτυχία σε προσωπικό επίπεδο, επαγγελματικό, οικογενειακό και ελπίζω αυτή εδώ η συνεδρίαση να είναι επιτυχής ε, σε σχέση με τους συμφωνισμούς που έχουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, να υπενθυμίσω τους, τις ομιλήτρες, ομιλητές ότι έχουμε ένα περιορισμό. Τρία είναι τα λεπτά και για να μπορέσουν να μιλήσουν όσο δυνατόν περισσότεροι. Τώρα, να δούμε τη Ρουμανία. Σίλα Μαλία Πέτερ έχει το λόγο. Είναι από τη Ρουμανία. Παρακαλώ. Doamna președintă, doamnelor și domnilor, în România, unul dintre domeniile... Proedre. Η România, είναι μια από τις χώρες όπου δεν υπάρχει καμία ισορροπία ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες στην πολιτική και το δυναμικό των γυναικών δεν χρησιμοποιείται λόγω διακρίσεων. Δεν υπάρχουν ούτε καν σχετικές νομοθεσίες. Η κατάσταση των γυναικών έχει βελτιωθεί την τελευταία δεκαετία, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ανισότητες. Τα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών όσον αφορά τη συμμετοχή στην πολιτική, στα όργανα λήψη αποφάσεων. Προχωράνε πολύ αργά. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι σε μια κοινωνία όπου οι γυναίκες έχουν πρόσβαση στην παιδεία και στα ίσα δικαιώματα, η πρόσβασή τους στην πολιτική ή και σε οποιοδήποτε άλλο τομέα δεν θα έπρεπε να παρεμποδίζεται. Αν δούμε όμως την εκπροσώπηση των γυναικών στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο, θα διαπιστώσουμε ότι από τους 333 βουλευτές, μόνο 37 είναι γυναίκες που εκλέγονται με το σταυρό. Και από τους γερουσιαστές, μόνο 8 είναι γυναίκες από τους 130. Ε, Βέβαια, είναι χαρά μας που πρώτη φορά έχουμε γυναίκα πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Οι γυναίκες, ωστόσο, γενικά είναι μόνο το 10,3%, ακόμα και μετά τις τελευταίες εκλογές του 2008. Είμαστε πολύ κάτω από το μέσο όρο, τον παγκόσμιο μέσο όρο, που είναι 15% και πολύ κάτω από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και τις χώρες ΩΣΑ. Επίσης, πολύ κάτω από το 37% εκπροσώπηση στις σκανδιναβικές ε, χώρες. Γνωρίζουμε πως η Σουηδία έχει το, ανώτατο, το, το ανώτερο ποσοστό του 43%. Αν κανείς κοιτάξει ρεαλιστικά την ισόρροπη εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στην πολιτική, θα πρέπει να λάβει υπόψη όλους τους συμμετέχοντες στην πολιτική ζωή. Λίγες γυναίκες δεν μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, ακόμα και αν οι δράσεις τους, η ενέργειά τους, η δουλειά τους είναι ψηλής ποιότητας. Ο λόγος πίσω από την χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο είναι ο εξής. Υπάρχει παραδοσιακή προκατάληψη για τους ρόλους των ανδρών και των γυναικών στην κοινωνία. Οι πολίτες αρνούνται να δουν τις γυναίκες ως πολιτικούς. Πιστεύουν ότι οι γυναίκες πρέπει να κερδίσουν κατά κάποιο τρόπο αυτό το προνόμιο. Δεν υπάρχει στήριξη λοιπόν, αλλά ούτε και κατάλληλη νομοθεσία. Μέσω της δικής μου δραστηριότητας ως βουλευτή και ως γραμματέος της Επιτροπής για τις Ίσες Ευκαιρίες στο Κοινοβουλίο μας, βασικός μου στόχος είναι να τροποποιήσουμε την υφιστάμενη νομοθεσία, την ισχύουσα νομοθεσία ή να φτιάξουμε και καινούρια έτσι ώστε να μπορέσουν οι γυναίκες να έχουν τα ίσα δικαιώματα, τα ίσα θεμελιώδη δικαιώματα με τους άνδρες. Θεωρητικά, οι άνδρες θα μπορούσαν και αυτοί να υποστηρίξουν τις γυναίκες. Αν και το πιο σύνηθες είναι οι γυναίκες να στηρίζουν τα δικά τους συμφέροντα και να προσπαθούν να βρουν λύσεις στα προβλήματά τους. Γι' αυτό και πιστεύω πως οι γυναίκες θα πρέπει να υψώσουν τη φωνή τους και να υποστηρίξουν τα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ. Και συνεχίζουμε την Κύπρο. Στην Κριστίνα Χελίδου έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, η Κύπρος έχει χαμηλή εκπροσώπηση γυναικών ε, στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στην πολιτική ζωή. Στην παρούσα σύνθεση της Βουλής θα πω μόνο ότι κυμαίνεται η εκπροσώπηση από 11% μέχρι 16% και αυτή η διακύμανση οφείλεται σε μετακινήσεις βουλευτών που κατέλαβαν τελικά άλλα αξιώματα ή εκπροσώπησαν την Κύπρο στο Ευρωκοινοβούλιο. Ε, δεν θα δώσω άλλα στοιχεία στατιστικά γιατί θα ήθελα, επειδή ακούστηκαν πολλά, να δώσω κατά την άποψή μου τις προτεραιότητες που πρέπει να έχουμε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο εθνικό επίπεδο αν είναι να προχωρήσουμε ε, σε γρήγορες γρηγορότερες τουλάχιστον αλλαγές ε, στα θέματα της ισότητας που θα φέρουν την πρόοδο τη σημαντική. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη προτεραιότητα είναι σίγουρα μια σφαιρική, συνεχής και εντατική προσπάθεια με πολιτικές σχέδια δράσης ε, και μέτρα συγκεκριμένα για καταπολέμηση των, των στερεότυπων ε, των φύλων και των στερεότυπων ρόλων των δύο φίλων στην οικογένεια και στην κοινωνία. Αν δεν γίνει αυτό, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ούτε στις αλλαγές στα κόμματα, που είναι η δεύτερη προτεραιότητα, πιστεύω, ε, που έχουν να κάνουν με αλλαγή νοοτροπιών, με τις εσωτερικές διαδικασίες των κομμάτων, με την, με την υιοθέτηση φιλικών, πιο φιλικών πολιτικών στην οικογένεια θέλει, όχι στο, στη γυναίκα, αλλά στην οικογένεια, σε σχέση με τις οικογενειακές υποχρεώσεις, τη φύλαξη των παιδιών, τη φύλαξη όσων έχουν ανάγκη για φροντίδα. Ε, και σίγουρα τη δέσμευση στα κόμματα για να προχωρήσουν σε αυτό που λέμε women's empowerment, την ε, ενίσχυση της γυναίκας για να παρουσιάζεται, να γίνει αναγνωρίσιμη, να καταπολεμηθούν όλες οι προκαταλήψεις μέσα από την εμπλοκή της και τη στήριξη των κομμάτων. Ε, οι προκαταλήψεις που θέλουν τη γυναίκα μακριά από την πολιτική. Επίσης, η τρίτη προτεραιότητα, θα έλεγα, που είναι και εξίσου βασική, είναι η ύπαρξη υποδομών φύλαξη των παιδιών, που είναι ένας παραδοσιακός ρόλος της γυναίκας, της μητέρας, και άλλα μέτρα για, για ίση κατανομή των ευθυνών μέσα στην οικογένεια. Επίσης, σίγουρα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ίδια η γυναίκα ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει όλη την ένταση όλη την προσπάθεια που χρειάζεται για να αποδείξει τον εαυτό της κτίζοντας μια καριέρα επαγγελματική και παράλληλα μπαίνοντα στην πολιτική ζωή. Δύσκολο χρειάζεται ενθάρρυνση η γυναίκα και σίγουρα ενθάρρυνση πρέπει να γίνεται και μέσα από το γυναικείο κίνημα και στο επίπεδο των εθνικών και το ευρωπαϊκό. Μια κοινή δράση είναι επίσης πολύ σημαντική στο επίπεδο της Ευρώπης αλλά και των γυναικείων οργανώσεων της κάθε χώρας είναι καλά να καταγραφούν σωστές πρακτικές οι οποίες να είναι στοχευμένες στην ε, κάλυψη των ελλημάτων, στην, στην πρόθεση της επίλυσης των προβλημάτων που εμποδίζουν τη γυναίκα να καταλαμβάνει ε, τη θέση της ε, στην πολιτική και οικονομική ζωή και θα ήθελα να πω ότι για μένα οι ποσοστώσει προσωπικά είναι, έχουν σίγουρα έναν επικουρικό λόγο και ρόλο. Οι ποσοστώσει μπορεί να θεωρηθούν θετικά μέτρα, προαιρετικά ή και υποχρεωτικά. Αλλά δεν λύουν το πρόβλημα μόνες τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στην Ελλάδα. Η κυρία Παναγιώτα Ζούνι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί αυτή η πρώτη μου επίσκεψη εδώ που χτυπάει η καρδιά και η πολιτική σκέψη της Ευρώπης συμπίπτει με μια ωραία επέτειο. Συμπίπτει με ένα πολύ γυναικείο θέμα. Ε, θα μπορούσα να πω πολλά, δεν θα πω, ε, θα, κρατήσω λιγότερο χρόνο ακόμα και από τα τρία λεπτά, γιατί είμαστε προς το τέλος της ε, συζήτησης. εξάλλου τα πράγματα στην Ελλάδα τα παρουσίασε η συνάδελφος η κυρία Τσαρουχά πολύ καλά. Ε, εντάχει τριπλασιάστηκε η συμμετοχή μας τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά δεν είναι αρκετό. Θέλω μόνο να πιάσω το νήμα από εκεί που περίπου το άφησε η Κύπρος για τους ε, ρόλους και για τις προκαταλήψεις και για τα, τα στερεότυπα όπου ελέγχθηκε από πολλές συνομιλήτριες και να καταθέσω μια σκέψη που ίσως ακουστεί λίγο ανορθόδοξη αλλά δεν είναι. Εμείς εδώ μέσα έχουμε αναθρέψει παιδιά όλες που ή έχουν ήδη πάρει την εξουσία στα χέρια τους, είναι αυτή η γενιά ή σε πολύ λίγο χρόνο θα μετέχουν στα κέντρα λήψης απόφασης. Εάν έχουμε κάνει σωστά τη δουλειά μας, τα πράγματα είναι πολύ καλά. Σε πολύ λίγο χρόνο θα έχουμε την απόλυτη ισότητα 50-50 με αυτούς τους άντρες που αναθρέψαμε, μιας και η κοινωνία είναι ανδροκρατούμενη ακόμα. Ε, τι θέλω να πω με αυτό. Ότι ίσως μέσα στα μέτρα και στις προτάσεις μας και στην ανάγκη δικτύωσης και στην ανάγκη μεγαλύτερης επαφής των κοινοβουλίων, ίσως μέσα σε όλα αυτά τα μέτρα της κοινωνίας, σκεφτούμε ότι έχουμε και ένα εργαλείο έμεσο αλλά ουσιαστικό αυτό της ανατροφής των νεαρών ανδρών και γυναικών που είναι και θα είναι στα κέντρα λήψης απόφασης. Έχουμε ένα ουσιαστικό ρόλο έμεσο ως γυναίκες που ανατρέφουν τους πολίτες και τους πολιτικούς για να αλλάξουμε αυτή την εικόνα που βλέπουμε ότι καθυστερεί. Αυτή η σκέψη έχει αρχίσει να συνυπολογίζεται και να συζητιέται σε κάποιες από τις διεθνείς συναντήσεις για την ισότητα και ήθελα να σας την καταθέσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και συνεχίζουμε στην Ουγγαρία. Η κυρία Σάμπου έχει το λόγο. Και εγώ θα είμαι σύντομη. Ευχαριστώ γιατί περνάει η ώρα. Σύντομη ε, ενημέρωση για τα σχετικά δεδομένα στην Ουγγαρία. Ζωφερά είναι και εκεί τα πράγματα. Όχι μόνο ε, σε σχέση με τα παγκόσμια αλλά και τα ευρωπαϊκά. Μετά την αλλαγή του καθεστώτος, ο λόγος ανδρών γυναικών πολιτικών στην Ουγγαρία μειώθηκε, επιδεινώθηκε δηλαδή το 90, το 95 μάλλον, στην παγκόσμια κατάταξη είμαστε στην 43η θέση. Το 99 κατεβήκαμε στην 86η θέση και τώρα είμαστε στην 127η. Ε, μιλάνε οι αριθμοί. Δεν είναι καλή η εικόνα. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Στο Κοινοβούλιο το κόμμα μου που είναι οικολογικό είναι το μόνο που έχει ποσόστοση και στην ε, κοινοβουλευτική μας ομάδα έχουμε 30% γυναίκες να κάνουμε ας πούμε σύγκριση. 386 είναι οι εθνικοί βουλευτές. 34 από αυτούς είναι οι γυναίκες πολιτικοί. Λιγότερο δηλαδή από το 9%. Εκτός από το δικό μας κόμμα, τα άλλα 5 έχουν λιγότερο από 5%. Για την ποσόστοση να πω κάποια πράγματα. Εγώ είμαι υπέρ της ποσόστοσης όχι επειδή είναι κανένα καταπληκτικό μόνιμο εργαλείο, αλλά χρειάζεται προσώρας. Και για να απαντήσω στη Σλοβάκα συνάδελφο, θα μιλήσω λίγο για αυτό το φόβο αν είναι ε, αντιπαραγωγικός ή όχι. Εγώ θα ήθελα να πω ότι το αντίθετο ισχύει, ήταν πολύ παραγωγικό. Όλοι, όλες οι γυναίκες τα πήγαν πολύ καλά Δηλαδή ο φόβος πως είναι αντιπαραγωγικό το μέτρο. Όχι, οι εμπειρίες μας ήταν πολύ καλές και θετικές. Πρέπει να δούμε το, τις ποσοστώσεις ως μέσον επίσης, γιατί πολλές φορές προβάλλεται το επιχείρημα ε, της, της ε, ισορροπίας μεταξύ ε, επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής όταν πρόκειται για τις γυναίκες. Επίσης είναι διαφωτιστικό το γεγονός ότι από το Μάιο έχουμε νέα κυβέρνηση και είναι σημαδιακό ότι δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα. Από τις υφυπουργού μία μόνο υπάρχει. Μεταξύ των υφυπουργών υπάρχει η εντύπωση ότι ε, μπαίνουν όρια, ε, δηλαδή αποτρέπεται η είσοδος ε, σε αυτές τις υπουργικές, υφυπουργικές θέσεις της γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η σχέση περίπου 70-30 κατά μέσον όρο. Ε, νομίζω παγκοσμίω είναι υψηλότερο το ποσοστό. για την Ουγγαρία θα μπορούσα να πω ότι το πρόβλημα είναι κοινωνικό, χρειάζεται καλύτερη ενημέρωση. Το 1997 έγινε μια συζήτηση για τις ποσοστώσεις και κατέστη σαφές ότι δεν ήταν γνωστό το θέμα αυτό. Η προβληματική των ποσοστώσεων δεν απασχολούσε ούτε την κοινή γνώμη ούτε τους πολιτικούς. Οπότε εκεί πολλά μπορούν να γίνουν ούτως ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη αφύπνιση, καλύτερη ενημέρωση Προσωρινό είναι το μέσο των ποσοστώσεων, δεν είναι μόνιμο, δεν είναι ο σκοπός, ούτε αυτός ο σκοπός είναι οι ποσοστώσεις, είναι ένα μέσον. Ε, εκτίμησα πολύ μια προηγούμενη παρέμβαση για τις μητέρες και τις άγαμες ε, γυναίκες ε, και εγώ είμαι μία από αυτές ε, υπάρχουν ορισμένοι εκπρόσωποι μας και χάρη στο κόμμα μου μπόρεσα εγώ να βρω μια ισορροπία μεταξύ δουλειάς και ζωής μου ε, οικογενειακής. Όχι λόγω του κράτους, όχι χάρη στην κυβέρνηση. Το κόμμα μου με βοήθησε. Ελπίζω λοιπόν ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμεθα πάνω σε αυτό το θέμα βελτιώνοντας ε, και ενισχύοντας την ενημέρωση πάνω σε αυτά τα θέματα συνδυασμού σταδιοδρομίας και οικογένειας και συμφωνώ με την Κυπρία συνάδελφο εδώ που υπογράμισε ότι δεν μιλάμε μόνο για το ρόλο των γυναικών ε, στην πολιτική. Πρέπει να εισαγάγουμε και πολιτικές φιλικές στην οικογένεια. Αυτό είναι ένα θέμα κλειδί. Και βέβαια στην Ουγγαρία πολλές γυναίκες ξαναγυρίζουν στην αγορά εργασίας αφού κάνουν τα παιδιά τους και αφού έχουν χάσει πολλές ευκαιρίες και αφού έχουν δει να συρρυκνώνονται οι προοπτικές. Ένα καλό στην Ουγγαρία είναι ότι το Κοινοβούλιο χάρη σε δική μας πρωτοβουλία όρισε έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο υπεύθυνο για ε, θέματα ε, επικούρησης των γυναικών που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας και εδώ θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω βέλτιστες πρακτικές για το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Συνεχίζουμε με το Μαυροβούνι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων των υποψηφίων χωρών ως εκπρόσωπος υποψήφιας χώρας. Ε, είναι μεγάλη μου τιμή που μου δίνεται η ευκαιρία να σας απευθύνω το λόγο ε, εξ ονόματος Επιτροπής Ισότητας Γυναικών από το Μαυροβούνιο ε, κατά την επέτειο αυτή των γυναικών. Πολλά έχουν επιτευχθεί, αλλά ακόμα πολλές δραστηριότητες έχουμε να ολοκληρώσουμε, ε, κυρίως εμείς οι υποψήφιες χώρες για να πραγματοποιηθούν τα δικαιώματα των γυναικών σε αυτό το τομέα. Σημαντικά θέματα ε, ε, συζητούνται στα Εθνικά Κοινοβούλια και στο Μαυροβούνιο θα ήθελα να παρουσιάσω την κατάσταση και την πρόοδο που επιτύχαμε σε αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το, στο Σύνταγμα προβλέπεται η αρχή απαγόρευσης διακρίσεων για οποιοδήποτε λόγο και στο άρθρο 18 λέει ρητά ότι υποχρεούται το κράτος να διασφαλίσει την ισότητα ανδρών και γυναικών και να αναπτύξει πολιτική ίσων ευκαιριών. Το 2007 το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου ε, υιοθέτησε τον νόμο για την ισότητα που ε, υποχρεώνει την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο να εφαρμόσει τις αρχές της ε, ισότητας των φύλων κατά την άσκηση της εξουσίας και να φροντίζει για ισορροπημένη εκπροσώπηση ε, σε διάφορες αντιπροσωπείες, ομάδες εργασίας κλπ. Όλα τα κόμματα θα πρέπει να φροντίζουν για το ίδιο όταν καταρτίζουν ψηφοδέλτια ή υποψηφίου ή υποδιορισμών ε, προσωπικότητες σε όλα τα επίπεδα, στις νομοθετικές δραστηριότητες, στο έργο των Επιτροπών, το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου. Δημιουργεί λύσεις ε, που αφορούν μέτρα μηχανισμούς επίτευξης της ισότητας των φύλων και κατάργησης των διακρίσεων λόγω φύλου. Κρίνοντας από το έργο του και τις αποφάσεις που ήδη έχουν εγκριθεί, το Κοινοβούλιο ακόμα δεν έχει αναπτύξει το δυναμικό που υπάρχει ικανοποιητικά. Η παρούσα κατάσταση έδειξε ότι οι γυναίκες ακόμη έχουν μικρότερη παρουσία στην πολιτική και αυτό είναι από τα μεγαλύτερα προσκόμματα για την άσκηση των δικαιωμάτων των γυναικών. Ε, 12,3% είναι οι γυναίκες στο κοινοβούλιο, που, είναι, που σε σύγκριση με τις άλλες χώρες είναι χαμηλό. Ο, ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος στο κοινοβούλιο είναι άνδρες. Από 11 επιτροπές μόνιμες μόνο δύο έχουν προέδρους γυναίκες. Τα τοπικά κοινοβούλια είναι παρόμοια στη σύνθεση και μία δήμαρχος υπάρχει ε, γυναίκα σε 21 δήμους. Υπάρχει μία μόνο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι υπουργό Επιστημών και η κατάσταση είναι παρόμοια και σε άλλα σώματα της κυβέρνησης. Μόνο στο δικαστική εξουσία είναι περισσότερες οι γυναίκες σας. Ε, οι κύριοι δικαστές, οι εισαγγελίσει, είναι γυναίκες Τώρα να θεωρείται ο εκλογικός νόμος για να βελτιώσει την εκπροσώπηση των γυναικών. Ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί, αν και οι ε, εκπρόσωποι του κόμματος πλειοψηφίας και της αξιωματικής αντιπολίτευσης ε, και οι δύο υπέβαλαν παρόμοιες προτάσεις για ποσόστοση στα ψηφοδέλτια και μετά στα αντιπροσωπευτικά σώματα στο τέλος της Ιαρινής Συνόδου του Κοινοβουλίου θα συζητηθεί το θέμα, ελπίζω να δοθεί καλή λύση. Η Επιτροπή Ισότητας παρακολούθησε το νόμο για την ισότητα ε, καθ' όλη την πορεία του. Τα ερευνητικά αποτελέσματα θα παρουσιαστούν αυτό το μήνα. Στο επίπεδο των πολιτικών κομμάτων υπάρχουν προγράμματα και μέτρα που στοχεύουν σε μεγαλύτερη εκπροσώπηση γυναικών, αλλά ο ρυθμός της εφαρμογή των μέτρων δεν ικανοποιεί. Πρόσφατα έγινε κάτι ελπιδοφόρο και ενθαρρυντικό. Δηλαδή το, η αξιωματική αντιπολίτευση ε, δέχτηκε τις ε, ποσοστώσεις και τις εφήρμοσε στην εκλογή εκπροσώπων, ε, αντιπροσώπων του, για το συνέδριο του κόμματος. Έτσι πιστεύουμε ότι πολλά ε, ακόμη μέλλον να γίνουν τόσο ώστε να υπάρχει καταστατική ισότητα στο, στο Μαυροβούνιο. Και τώρα ο λόγος στην κυρία Μερόκα, ε, μέλος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε και κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ για την πολύ ζωντανή συζήτηση. Η Επιτροπή του Κοινοβουλίου τα τελευταία 6 χρόνια από τότε που εγώ είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής δηλαδή, ε, θίγει αυτά τα θέματα διαρκώς ε, προς την Κομισιόν και προκαλεί το Συμβούλιο στο να λάβει αποφάσεις. Ε, δύο μέρες μόλις πριν είχαμε συνάντηση με την Επίτροπο, την κυρία Ρέντινγκ, για το θέμα αυτό και με χαρά ακούσαμε ότι όχι μόνο στον πολιτικό τομέα αλλά και στον επιχειρηματικό τομέα σε επίπεδο δηλαδή τραπεζών υπάρχει μεγάλο ζήτημα για την αλλαγή αυτής της, της ισορροπίας μεταξύ των φύλων και αυτά που μας είπε για τη στρατηγική της προς αυτό το τομέα είναι ότι όλο αυτό το έτος ε, η Κομισιόν θα δει πώς μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα στην Γενικό Συμβούλιο, στο Διοικητικό Συμβούλιο μάλλον των επιχειρήσεων και σε ένα χρόνο θα μιλήσει λοιπόν για ποσοστώσεις. Ε, θα το δούμε και στην πολιτική, το έχουμε δει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπήρξε μεγάλη ε, αύξηση πολιτικών, γυναικών ε, πολιτικών γυναικών. Ξέρουμε πως δεν είναι ικανοποιητικό το, πρά, το, το επίπεδο στο οποίο έχουμε φτάσει τώρα, πάντως... Ε, έχουμε την έκθεση της Σιβώνα Πλάμ που μιλάει για τις γυναίκες πολιτικούς στην Ευρώπη και την κατάσταση ισότητας ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες για το 2010. Κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων κατέστη σαφές ότι αυτό για το οποίο μιλάμε σήμερα είναι ότι βασικά οι γυναίκες ε, βγαίνουν από, ε, έχουν μάλλον ε, καλή εκπαίδευση. Ναι, στην οικονομία δεν έχουμε αρκετές γυναίκες. Έχουμε αρκετές γυναίκες στη πανεπιστήμια, στις, στην κοινωνική πρόνοια αλλά είναι περισσότερο οι πολιτικές και οι οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη Οι γνώσει αυτών των γυναικών που προέρχονται πραγματικά από τη βάση θα έπρεπε να είναι πολύ σημαντικό. Σημαντική και χρήσιμη. Εδώ, ας πούμε, στο Κοινοβούλιο θα έπρεπε να υπάρχουν αναλογικά 10 ε, ε, ευρωβουλευτίνες ε, Ρωμά. Αλλά υπάρχει μόνο εγώ, μία. Και δεν ξέρω πόσες γυναίκες μπόρεσαν να βγουν από τέτοιες καταστάσεις που έχουν υποστεί μεγάλες ε, ε, διακρίσεις. Έχουμε ε, ανήπαντρες γυναίκες που έχουν υποστεί άλλες φιλετικές διακρίσεις και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τις δυνατότητές μας ως γυναίκες ηγέτες, ώστε να εξασφαλίσουμε πως από το βάση θα προέρχουν νέες γυναίκες από οποιοδήποτε υπόβαθρο, από οποιοδήποτε κατάσταση, ακόμα και όταν είναι πιο δύσκολη η κατάσταση, γιατί οι πολλαπλές διακρίσεις μπορεί να είναι ακόμα πιο ε, να καταστούν ακόμα πιο δύσκολη την πορεία του στην πολιτική. Και αυτό τόσο για την πολιτική ζωή όσο και για την επιχειρηματική ζωή. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω από όλους σας τα Εθνικά Κοινοβούλια να στηρίξετε την Επιτροπή των Γυναικών και στα κόμματά σας επίσης. Ώστε όλοι όσους εκπροσωπείτε να έχουν τη δυνατότητα πέρα από σας και ίσως και πάνω από σας να φτάσουν σε θέσεις από όπου να μπορούν πραγματικά να οδηγήσουν σε αλλαγή. Και για αυτό το στόχο η Επιτροπή των Γυναικών μπορεί να χρησιμεύσει. Κυρία Ρόμπινσον. Uh, Σας ευχαριστώ. Έχω πολύ λίγο χρόνο, αλλά θέλω μόνο να πω πως πραγματικά ήταν ε, διαφέρουσα η συζήτηση. Και ως πρεσβύτερη με εντυπωσίασαν κάποιες πολύ ε, ικανές και φράδες ε, νεαρές γυναίκες. Να σας πω όμως ότι 17 κοινοβούλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μόλις 27 γυναίκες μέλη. Ε, θα πρέπει να το σκεφτούμε στις χώρες μας, στο πλαίσιο της κάθε χώρας, ε, πώς θα οδηγηθούμε σε αλλαγές. Και αυτό είναι στο οποίο εγώ παροτρύνω. Ίσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να δώσει ένα μήνυμα ότι θα πρέπει να δοθεί επιγόντως προσοχή στις χώρες όπου υπάρχουν λιγότερο από 25% εκπροσώπηση γυναικών στο Κοινοβούλιο, ώστε να ενθαρρύνει την κατάσταση γιατί το ποσοστό είναι ψηλότερο εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Και γιατί είναι αυτό σημαντικό, γιατί υπάρχει μια κρίσιμη μάζα γυναικών στο κοινοβούλιο, τότε μπορείς να ασχοληθείς με διάφορα θέματα. Δηλαδή, περισσότερες γυναίκες στην οικονομική κρίση, γυναίκες περιθωριοποιημένες που χρειάζεται να ακουστεί η ζωή τους, όλα αυτά τα θέματα. Και να φτιάξεις και τις ιεραρχήσεις τις προτεραιότητες. 25% είναι η μίνιμουμ κρίσιμη μάζα σε ένα σύγχρονο κοινοβούλιο, κατά τη γνώμη μου. Πολλά κοινοβούλια λοιπόν είναι πολύ κάτω από αυτό το ποσοστό και το δικό μου. Και αυτό είναι θέμα επίγουσες ανάγκες και μπορούμε νομίζω να ενθαρρύνουμε με τους ΔΕ για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε πραγματικές βαθιές αλλαγές. Ευχαριστώ. κυρία Φοντέν παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ σύντομη θα είμαι για να πω, να σας συγχαρώ μάλλον που πήρατε αυτή την πρωτοβουλία. Εγώ θεωρώ ότι ο διάλογος εδώ ήταν πολύ δυνατός, ενδιαφέρον, επικοδημητικός μάλιστα. Και είναι σημαντικό γιατί αυτό μάλλον επιθυμούσατε. Να επανέλθω απλώ σε ένα θέμα το οποίο αναφέρθηκε. Το περίφημο θέμα των ποσοστώσεων. Σίγουρα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Εγώ θα έλεγα περισσότερο θα χρησιμοποιήσω τον όρο ισότητα, όχι ποσόστοση. Ισότητα. Ε, ίσες ευκαιρίες. Είναι πολύ πιο καλός όρος. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε εξάλλου. Για λόγους ε, δικαιοσύνης, δημοκρατίας. Μην το ξεχνάμε. Και για τον ίδιο λόγο που δεν ζητάμε κάτι που να είναι ε, υπέρ μας. Ε, υπήρχε το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις ασφάλειες όπου η, ακούστηκε ότι οι ασφαλιστές λέγανε ότι οι γυναίκες οδηγούν καλύτερα από τους άνδρες και κάτι τέτοια πράγματα. Αυτό δεν το θεωρώ σωστό. Ούτε τέτοια θετική διάκριση θέλω. Ισότητα. Ισότητα τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Επίσης αναφέρθηκε το τι έχει γίνει στη Γαλλία σε επίπεδο ε, δημοτικών εκλογών και εδώ είναι κάτι σημαντικό. Εγώ έχω πολλές επαφές σίγουρα με δημάρχους, άντρες όπου είδα ότι ήταν, είχαν μια επιφύλαξη πριν κατά το παρελθόν ε, διστακτική, καχύποπτα και σήμερα τι λένε ότι μπο, ωραία είχαμε μια εξέλιξη πάρα πολύ θετική και θεωρούν ότι η αλλαγή ήταν ε, προς το καλύτερο όχι μόνο για τα, τη δημοκρατική πτυχή αλλά και για τους πολίτες λοιπόν ισότητα ε, ανδρών γυναικών σε επίπεδο δημοτικών συμβουλίων είναι κάτι το οποίο είναι θετικό και θεωρώ ότι ε, το είδαν και οι άντρες σαν κάτι σημαντικό. Έχουμε την πραγματικότητα αυτής της ισότητας που δείχνει τις θετικές πτυχές και όλοι αναγνωρίζουν ότι οι γυναίκες ισότιμες στα δημοτικά συμβούλια συνέβαλαν τα μέγιστα και θεωρώ ότι εδώ έχουμε δηλαδή τον πυρήνα από όπου θα ξεκινήσει μια εξέλιξη όχι με μια μαϊκή ράβδο σιγά σιγά που θα δώσει καρπούς. Φυσικά αυτό συνοδευόμενο με μια κινητοποίηση όπως αναφέρεται και εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λόμπι των Γυναικών. Ε, μπράβο πάλι, ξανά να σας πω κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε έτσι. Και η κυρία Πιέτη Κάινεν ε, έκανε ε, κάτι πολύ καλό με τις προτάσεις της. Θα εμπλουτίσουν ε, σίγουρα όλες αυτές οι απόψεις εδώ μέσα την έκθεσή της. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Πιετικάινα θα πάρει το λόγο για να κλείσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τα πολύτιμα σχόλιά σας και τις ιδέες σας για την εκθεσή μου που προετοιμάζω και για την ευαισθησία που είχατε να μας αναφέρετε την κατάσταση πως έχει στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Να αναφέρω τα εξή. Καταρχήν, ναι, θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε τι είδους ε, εστιασμένες δράσεις θα μπορούσαμε να κάνουμε στα κράτη-μέλη όπου τα νούμερα είναι χαμηλά σε συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Δεύτερον, το ρόλο της παιδείας όπου δηλαδή θα μπορούσαμε να δούμε νέα κορίτσια και να τους δείξουμε ότι η πολιτική ταιριάζει με τις γυναίκες. Και έπειτα να δούμε και τη κοινωνική διάσταση. Επίσης, ε, ήταν πολύ ωραία αυτή η σημερινή συνεδρίαση και σίγουρα θα είμαστε σε επαφή και στο μέλλον θα προσπαθήσουμε να συγκεκριμενοποιήσουμε τις δράσεις μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και με αυτό να ευχαριστήσω όλους όσοι πήραν ή όσες πήραν το λόγο για ένα επικοδομητικό διάλογο. Επίσης να επενθυμίσω και άλλα σημαντικά θέματα σε σχέση με την Διεθνή ημέρα της γυναίκας στο Στρασβούργο και, στο Βρυξελ, και στις Βρυξέλλες ε, συνολομέλεια στο Στρασβούργο Φέρυπιν μαζί με την ε, Επιτροπή και την ε, Ουγγρική Προεδρία θα εορταστεί πανηγυρικά αυτή η μέρα επίσης σεμινάρια για δημοσιογράφους για, με το θέμα η γυναίκα σε ηγετική θέση Επίσης οργανώνεται ένα σεμινάριο για τον αγώνα 100 χρόνων της γυναίκας ε, και η Γκουε οργανώνει μία διάσκεψη. Ε, επίσης οι πράσινοι έχουν ένα θέμα σήμερα το οποίο ασχολείται με τα θέματα των γυναικών. Εγώ θεωρώ ότι σήμερα, μάλλον δείξαμε σήμερα ε, τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, ποια ήταν η πρόοδος, αλλά και ποιες είναι οι προκλήσεις για το μέλλον. Θεωρώ ότι μαζί, από κοινού και με τα ΜΜΕ θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τα θέματά μας και να δείξουμε ότι όλοι θέλουμε, όλοι μπορούμε, ότι μπορούμε από κοινού να κάνουμε αυτόν τον αγώνα για την ισότητα. Είμαι πεπισμένη ότι θα πετύχουμε με τους στόχους μας και πρέπει να δείξουμε ότι δεν δεν είμαστε διατεθειμένες να περιμένουμε άλλα 100 χρόνια για να δούμε μια καλύτερη κοινωνία. Θέλουμε μια ισότιμη κοινωνία ανδρών, γυναικών και παιδιών. Ευχαριστώ όλους και όλες που ήταν παρόντες σήμερα. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και ένα κόκτελ, ένα ποτό, ένα όροφο κάτω, εδώ σε αυτό το ίδιο το Και να κλείσω λέγοντας ξανά να ευχαριστώ στους συμμετέχοντες, στην Γραμματεία για την Ισότητα που δούλεψε με αυτό εδώ το θέμα. Ευχαριστώ και τους Γερμινείς. Συγγνώμη ε, ότι πάλι τους κλέψαμε λίγα λεπτά, αλλά ε, ε, τους ευχαριστούμε. Όλοι ε, είσαστε εκπρόσεκτοι στο ποτό. Ευχαριστώ.